Συνάδελφοι, καλημέρα. Ας ε, ξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ πέρα δύο μεγάλα θέματα. Δύο σκέλη του τραπεζικού πακέτου τα οποία είναι στη φάση των ε, τροπολογιών. Ε, πολλή δουλειά βεβαίω έχουμε. Λογικό. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως. Δεν θα πω τίποτα. Θα δώσω τον λόγο στον Γκουινάρ Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ τους κοιόδες εισηγητές ε, και τους άλλους ε, βουλευτές. Υπάρχουν γύρω στις 600 ε, τροπολογίες που όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε ήταν αναμενόμενο. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια βασικά πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν οι τα κεφαλαιοποιημένα ιδρύματα από επιπλέον απαιτήσει κεφαλαιοποίησης ε, αν ε, μια τράπεζα είναι ήδη απαρκώς κεφαλαιοποιημένη αυτό πρέπει να επηρεάσει και το επίπεδο των απαιτήσεων ε, κεφαλαιοποίησης και απορροφήσεις ε, ζημιών. Επίσης ε, θα πρέπει το επίπεδο του ε, χρέους βεβαίω να ληφθεί υπόψη σε σχέση με το τίλα. Και τρίτον η αναλογικότητα στην οποία δεν θα επιμείνω αλλά βασικό κομμάτι είναι ότι οι τράπεζες οι οποίες δεν θα πηγαίνουν προς ε, διάσωση δεν χρειάζεται να έχουν αυτές τις ε, ικανότητες απορρόφησης ε, ζημιών. Μπορούν απλά να ρευστοποιηθούν. Και βεβαίως ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά επίμαχο είναι η συζήτηση περί ενός μορατόριου όπου είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και εγώ στην έκθεσή μου είχα πει ότι για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ενός πολύ μακροχρόνιου μορατόριου μπορεί τελικά η εγχείρηση να πετύχει αλλά ο ασθενής να πεθάνει δηλαδή η τράπεζα στην πραγματικότητα να μην ανακάμψει και όσον αφορά τις ε, τροπολογίες που εστιάζουν ε, κυρίως σε αυτά το ε, αρμοδιότητες ε, περί ενός μορατόριου πρόοδου της ε, διάσωσης. Πολλοί σκιώδεις συγητές και συνάδελφοι λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα μορατόριο, άλλοι ότι θα πρέπει να είναι μόνο στη φάση της διάσωσης. Εγώ εκτιμώ ότι πολύ εύκολο νομίζω σχετικά εύκολο να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις Όσον αφορά την επιλεξιμότητα και το ύψος ε, των ε, απαραίτητων αυτών αποθεματικών ε, και το ζήτημα της αδιακής κατάληξης δεν πρότεινα εγώ κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ως όριο και ήταν συνειδητή απόφαση και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συντονίσουμε εδώ πέρα αυτό το θέμα με το θέμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων του σχετικού κανονισμού. Λοιπόν... Και Όσον αφορά το αποθεματικό για την απορρόφηση ζημιών, εντάξει θα μπορούσαμε ίσως να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα για τις ελάχιστες αυτές τις απαιτήσεις πάνω από το επίπεδο τηλεπτή θα τα αναπτύξω αυτά περαιτέρω και αναμένω να καταλήξουμε σε κάποιους ε, συμβιβασμούς. Το θέμα λοιπόν ε, της ε, κατεύθυνσης που θα δοθεί πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να έχουμε κάποια κατεύθυνση και να πάμε προς, προς τα εκεί να δούμε τώρα τι θα προκύψει από τις συζητήσεις και τώρα όσον αφορά τα εσωτερικά αυτά αποθεματικά απορρόφησης ζημιών που είναι ίσως το πιο περίπλοκο ζήτημα γιατί έχουμε χώρες προέλευσης ε, και χώρες οι οποίες ε, φιλοξενούν υποκαταστήματα. Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοια εσωτερικά αποθεματικά στην Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Άλλοι λένε ότι θα πρέπει να το δούμε στην Τραπεζική Ένωση. Θεωρώ ότι στην πραγματικότητα οι απαιτήσει για τις τράπεζες είναι κάπως πιο α, σοβαρές. Ας ακολουθήσουμε αυτό το σκεπτικό και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα πρέπει να επιτύχουμε, να διατηρήσουμε την ισορροπία που είχαμε πετύχει στην σχετική οδηγία. Θα προκύψουν βεβαίω και άλλα ζητήματα. να προσθέσω μόνο το εξή. Κάποιοι συνάδελφοι επίση ε, έστειλαν και τροπολογίε που στόχο έχουν να ανοίξουν ε, ξανά την όλη συζήτηση και ε, διστάζω να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή είμαι αντίθετος. Δεν είναι τώρα η ώρα να ξεκινήσουμε τέτοια συζήτηση. Λοιπόν, αυτά και ευχαριστώ να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων και μετά θα περάσουμε στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για αυτά τα σημεία που θίξατε. Ήδη έχω επενθυμίσει πρέπει να πω στους συναδέλφους Πρόκειται για μία άσκηση να προσπαθούμε να συνθέσουμε αντίθετες απόψεις κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα έναν ζωντανό διάλογο αλλά πιστεύω ότι είναι ρεαλιστική η θέση του εισηγητή ο κύριος Σίλβα Περέιρα έχει το λόγο Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον εισηγητή Συζητήσουμε, συνεχίζουμε λοιπόν την ε, συζήτησή μας και τις προτάσεις μας για τον μηχανισμό διάσωσης των τραπεζών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συζήτηση σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα. Στόχος βεβαίως είναι να ενσωματωθούν τα διεθνή standards σε ό,τι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση. στα υπάρχοντα standards που έχουμε για τις ελάχιστες απαιτήσει. Αυτό από τη φύση του είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό ζήτημα, ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα. Αλλά αυτή η τεχνική ορολογία έχει πολύ συγκεκριμένα σημεία που φύγονται σε ό,τι αφορά τι τράπεζε αλλά και του πολίτε. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο σύστημα σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, αλλά και ένα αξιόπιστο πλαίσιο για τις δύσκολες στιγμές που μπορεί και να έρθουν. Και όταν αυτές οι δύσκολες στιγμές έρθουν, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε τις επενδύσεις αλλά και τις καταθέσεις των πολιτών. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους και τον εισηγητή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κοινά σημεία και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, γρηγορότερα. Όπως ε, πολλοί συνάδελφοι, 600 περίπου προτάσεις για τροπολογίες έχουμε. Σε κάποια σημεία οι τροπολογίες παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές θέσεις. Σε κάποια άλλα σημεία είναι συγγενείς με τις θέσεις του εισηγητή. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην τροπολογία που αφορά την ε, προδιάσωση κατάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν έχουμε πρόταση διαγραφών. Αυτή είναι η θέση της δικής μας πολιτικής ομάδας. Σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε και τελείως διαφορετικές θέσεις σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την δυνατότητα πρόσβαση στο MRL. Έχουμε, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τα MRLs. Και προέκυψαν αρκετά ζητήματα ε, να σκεφτούμε συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας σε ό,τι αφορά την διαγραφή οποιασδήποτε κατευθυντήριας πρότασης. Θέλω εγώ τώρα να επικεντρωθώ στις δικές μας προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για τα MRLs αλλά και τον συντονισμό αυτών των ελάχιστων επαιτήσεων είναι ανάγκη να ενδυναμωθεί η χρηματοπιστική σταθερότητα αλλά και τα MRL αυτά να προσφέρουν τη δυνατότητα επανακεφαλαιοποίησης της οικονομίας. Είναι ανάγκη λοιπόν να επανασυντονιστούν και τα πιστοτικά ιδρύματα να μην αναγκάζονται να προσφέρουν ελάχιστες απαιτήσει που δεν είναι αναλογίες με τις δυνατότητές τους. Πρέπει να υπολογιστούν τα MRL αυτά από τις αρμόδιες αρχές και να διασαφινιστούν στις νομικές προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε οντότητας και θα βρίσκονται στην ευχέρεια της κάθε αρχής. Συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα MRLs, κάτι το οποίο θα πρέπει να υπολογίσετε μετά την διάσωση και όχι πριν. Θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης, να λαμβάνουν υπόψη τους το αποθεματικό της κάθε τράπεζας. Δευτερευόντως, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τα MRL και την ε, συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια ομαλή διαδρομή μέχρι ε, την ε, συγκέντρωση των MRL αυτών, των ελάχιστων αυτών απαιτήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για παράδειγμα οι αρμόδιες αρχές να θέτουν μεγαλύτερες περιόδους για να μπορέσουν τα, τα ιδρύματα να συγκεντρώσουν τα χρήματα για, τις, ε, για αυτά τα MRL, για τις ελάχιστες αυτές απαιτήσει. Αυτή η μεταβατική περίοδος για τις τράπεζες θα μπορούσε να είναι μακρύτερη για ορισμένα ιδρύματα, για κάποιες τράπεζες για παράδειγμα, ακριβώς λόγω αυτής της αρχής αναλογικότητας. Όπως είπα είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι οι αγορές μπορούν να απορροφήσουν αυτά τα MRLs. Υπάρχουν, έχουμε πριν ανοιχτές τροπολογίες στα σημεία αυτά. Και ανυπομονώ, λοιπόν, για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας, από κοινού με τον εισηγητή στους επόμενους μήνες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία, να μπορέσουμε να συμβιβαστούμε και να έχουμε και θετικά αποτελέσματα πάντοτε προς όφελος της ε, χρηματικής σταθερότητας, της οικονομικής σταθερότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Περέιρα. Η κυρία, ο κύριος Καμάλ έχει το λόγο. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τους κοιόδης εισηγητές για αυτές τις ε, συζητήσεις. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που προτείναμε εμείς. Πρώτα, σε ό,τι αφορά την αρχή της ευελιξίας. Δευτερευόντως, την δυνατότητα να συμμορφώνονται τα MRL σε αυτά ανάλογα με το πιστοτικό ίδρυμα για το οποίο αναφερόμαστε. Και πάλι ευελιξία και επίσης σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα απορρόφησης των συνεπειών. Αναφέρομαι σε αυτό το μορατόριο. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μιλάμε για τα ζητήματα τα οποία πρέπει να θίγουμε. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω. Παραμένουμε αντίθετοι στις προληπτικές αυτές ενέργειες που προτάθηκαν από την Επιτροπή. Είμαστε διατεθειμένοι να δούμε την άλλη πλευρά, αλλά προς το παρόν θεωρούμε ότι είναι πιθανότατα επιζήμιες τέτοιου τύπου προληπτικές ενέργειες. Θέλουμε λοιπόν είτε να διαγραφεί τελείως το κομμάτι αυτό ή να βρούμε έναν συμβιβασμό σε ό,τι αφορά τώρα τα MRL θεωρούμε ότι η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι ε, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να είναι ευέλικτη και να συντονίζεται με τις δυνατότητες του κάθε συγκεκριμένου ιδρύματος. Διαφορετικά θεωρούμε ότι θα είναι επιζήμιο το αποτέλεσμα. Η αρχή διάσωσης θα πρέπει να μπορεί να ζητάει υψηλότερες ελάχιστες απαιτήσεις μόνο όταν το θεωρεί αναγκαίο. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, θεωρούμε και πάλι ότι θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της συγκεκριμένης αρχής να προσαρμόζεται. Θα πρέπει τα MRL αυτά να κινούνται μεταξύ 75 και 90 Αλλά η Επιτροπή έχει προτείνει MRL στις τάξεις στο 90%. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να κινούνται ανάμεσα στα ποσοστά αυτά και να αποφασίζουν ποιο ποσοστό αναλογεί σε κάθε επιχείρηση. Ακριβώς επειδή υπάρχουν διεθνή standards θα πρέπει και εμείς να συμβιβαστούμε. Τα διεθνή αυτά standards αναφέρονται σε 75-90% MRLs. Επομένως θα ήταν περίεργο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει αυτήν την ε, δυνατότητα κίνησης μεταξύ των δύο αυτών ποσοστών. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίζει τη θέση αυτή. Θεωρούμε τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 55, ότι η αρχή θα πρέπει να εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά η αρμόδια αρχή. Θα πρέπει η κάθε, με άλλα λόγια, θα πρέπει το κάθε πιστοτικό ίδρυμα να αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες και να μην είναι όλα στην αρμοδιότητα της εκάστοτε εποπτικής αρχής. Σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα, δεν στηρίζουμε κάποιες τροπολογίες που αναφέρονται στην επιλεξιμότητα. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάμπολα άλλα σημεία, αλλά αυτά είναι τα βασικά. Ε, και ανυπομονώ κι εγώ να συνεργαστώ με τους συζητητές. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο και τώρα είναι ο κύριο Κλίντσα. Θα μιλήσω για την άλλη, αλλά για τον κύριο Κορνίγια που δεν μπορούσε να έρθει. Και σα διαβάσω το κείμενο που εκείνο έχει ετοιμάσει. Πρώτα-πρώτα ευχαριστούμε τον Γκούνα Χέκμαρ και την γραμματεία. Ε, ήταν ε, παραγωγικές οι συναντήσεις και με την Τράπεζα και με την Κομισιόν και ε, με την Αρχή Τραπεζών ακριβώς Όπω και για τον SRB, είπαμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Τραπεζική Ένωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορετικέ ρυθμίσει για τα MRL. Και θα πρέπει να δούμε τι θα εξαιρείται από αυτές τις κεφαλαιολογικές απαιτήσει. Θα πρέπει να είναι ο κανόνας τα MRL και νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο δυνατό μέσο και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει πλήρη υπαγωγή για όλες τις τράπεζες. Και θέλουμε αυτό να είναι ένα από τα μέσα ούτως ώστε η στατική την εκαθάριση να λειτουργεί. Επομένως αυτό θα πρέπει να εξετάζεται τράπεζα. Αυτό προτιμώ, λέει ο κύριος Κορνιγέ. Πάντως και οι δύο προτινόμενες λύσεις είναι λογικές και όσον αφορά τα μορατόρια δεν βλέπω τι θα κερδίσουμε, αλλά θα πρέπει να συνεχιστούν οι επαφές με το, την SRB και το EBA όσο χρειάζεται. Όταν θεσπίζουν αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολυμορφία του τραπεζικού τομέα. Αυτό είναι κάτι το καλό. Και να μην ξεχνούμε ότι οι τραπεζές μας δρούν σε έναν ε, παγκοσμιοποιημένο κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ΚΟΕ. Μάρτιν Σίλντεβαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους συναδέλφους για την δουλειά που έκαναν. Ήδη στο παρελθόν το παρελθόν μου έχει πει πολλές φορές ότι αμφιβάλλουμε για το αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην πράξη μέσα όπως το MRL και το TILAC και θα θέλαμε να υπάρχει μια πολιτική εναλλακτική για να δείξουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διάσωση των, των τραπεζών με χρήματα των φορολογουμένων αλλά με διαφορετική λύση ειδικά για συστημικές ε, τράπεζες αλλά δεδομένων των πλειοψηφιών στο Κοινοβούλιο δεν ε, έχουμε προφανώς επιτύχει τον στόχο μας οπότε έχουμε επικεντρωθεί στο BRD και προσπαθούμε να περιορίσουμε ακριβώ την κοινωνικοποίηση των ζημιών. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 32 περί προληπτικής κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ περισσότερο γιατί είχαμε ακριβώς το μπέιλινος παραθυράκι που είχε χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς ζητάμε με την τροπολογία μας 196 να διαγραφή αυτό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 32 και αυτό το οποίο θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι η ρύθμιση του MRL αφορά βεβαίως και τις, ικανο... και τις αρμοδιότητες των ε, ρυθμιστικών αρχών και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις τροπολογίες 202 και 39 που αφορά τις μη ασφαλισμένες ε, καταθέσεις και θα πρέπει βεβαίως ε, και οι πιστωτές ε, σύμφωνα με το άρθρο 75 να αποζημιωθούν με δημόσια λεφτά. Οπωσδήποτε δεν μπορεί αυτό να είναι ένα επιτυχημένο καστό Μπέιλιν. Επιπλέον έχουμε τις τροπολογίες 206 και 216 που έχουμε υποβάλει για τα δομημένα προϊόντα στα οποία θα πρέπει να ενταχθεί το MRL τα πολύπλοκα αυτά μέσα και τα άλλα παράγωγα και τα λοιπά κατά την άποψή μας ε, δεν ενδείχνεται ιδιαίτερα για Μπέιλιν γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια κοινή θέση η οποία θα επανέρχεται στις προδιαγραφές που διατυπώνονται εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε επικριτικά το μέσο αυτό, αλλά θα πρέπει στην ε, πράξη να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και να μην περιορίζονται οι δυνατότητες μας στην περίπτωση διάσωσης ε, τραπεζών και ειδικά να περιοριστούμε στα άρθρα 45 C και D. Θα πρέπει λοιπόν οι διασώσεις ε, να έχουν μια νομική ασφάλεια και να μην περιορίζονται στις κινήσεις των εποπτικών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν πολύ περισσότερο να έχουν την διακριτική ευκαιρία να αποφασίζουν ποια μέσα θεωρούν οι ίδιες ε, σωστές όσον αφορά δε την κατεύθυνση του αποθεματικού αυτού το οποίο συζητείται σε διάφορα θεσμικά όργανα όπως ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Με θέσεις αρκετά κοντά στις ε, δικές μας έχουμε την οδηγία περί κεφαλιακών απαιτήσεων και στο άρθρο 45ε. Το βλέπουμε πολύ επικριτικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ πέρα από, σκληρές από πολύ σκληρές ποσοστώσεις και ύψος αυτών των αποθεματικών πηγαίνουμε περισσότερο προς την κατεύθυνση κάποιων συστάσεων. Γι' αυτό προτείνουμε στο άρθρο 384 στην τροπολογία 384 να διαγραφεί το, 200, το άρθρο 240 ε. Επίσης με αυτά τα οποία αναφέρει το άρθρο 55 ως υποχρεωτικές μπέιλιν για λαδαπούς επενδυτές είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χαιρετίζουμε. Όμως οι εξαιρέσεις της ε, παραγράφου 2 αφορούν περισσότερο ιδρύματα τα οποία δεν έχουν παγκόσμια συστημική σημασία. Αυτά για το BRD. Αναμένουμε και την περαιτέρω συζήτηση με τον εισηγητή και τους κοιότητες εισηγητές ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ θέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος Έρνης. Ουρτάσουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή για την καλή δουλειά του. Μια γενική σκέψη πρώτα-πρώτα. Πολύ κακή η κατάληξη αυτής της εντολής θα ήταν αφού μερικές ομάδες δεν θέλουν να συμβιβαστούν τότε ε, θα πρέπει να, να, απαντήσουμε ότι και για τα δύο θέματα ή θα συμβαστούμε ή για κανένα από τα δύο. Ε, πρέπει να βρούμε τελικά μια πλειοψηφία και γι' αυτό σας λέω για αυτό το πακέτο, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε κάποιο σχέδιο για τη διάσωση. Και οι τροπολογίες, πολλές από αυτές τουλάχιστον, που πολλές φορές δυσκολεύουν τις ε, αρχές διάσωσης, θα πρέπει να τις αποφύγουμε. Και όσον αφορά τη μέτρηση του MRL και λοιπά και για την αρχή τραπεζών, όλα αυτά τα είπαμε χτες, άρα για τον υπολογισμό του MRL δεν θα πρέπει να βάλουμε σε αυτόν τον υπολογισμό ένα, μια οροφή. Να έχουμε ένα κατόριο και μετά να δούμε οι αρμόδιες αρχές προς τα που θα πάνε. Επίσης και για τα, πάλι για τα MRL θα πρέπει να έχουν τέτοια ποιότητα που να βοηθούν στο Μπέιλιν. Και για την υπαγωγή υπάρχει μια τροπολογία που αν δεν κάνω λάθος αναφέρει ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται αυτές οι αρχές διάσωσης να έχουν ε, να, να, να ασχολούνται με στοιχεία του παθητικού πέραν του πρώτου πυλώνα. Αν θέλουν να πάνε στο δεύτερο πυλώνα όμως θα έπρεπε να τους επιτρέπεται λέω γιατί έτσι τις περιορίζουμε πάρα πολύ αυτές τις αρχές. Guidance τώρα. Χτες για την αρχή τραπεζών τα συζητήσαμε και για τον μηχανισμό SSM. Αν όμως έτσι περιορίσουμε την guidance και δεν καλύψουν το CBR με το MRL, ε, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ή θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση για τα MRL ή μάλλον αυστηρή προϋπόθεση για τα MRL και θα πρέπει να καλύψουμε το CBR στην guidance. Και για να έχει νόημα θα πρέπει να υπάρξουν για να έχει νόημα θα πρέπει να προβλέπονται και συνέπειες. Με κάποια άλλα θέματα τώρα όσον αφορά το μορατόριο ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα για τον SSM χθε. Ότι μορατόριο πριν την διάσωση δεν χρειάζεται σε, κάποια, σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Αποδείχθηκε ότι έτσι ίσχυσε στην υπόθεση Banco Popular και όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση θα πρέπει να υπάρχει περίοδος χάριτος στην οδηγία. Και αν βάλουμε, τη, αν βάλουμε πάντως και ρήτρα grandfathering και περίοδο χάριτος, αυτό παραπάει, είναι υπερβολικό. Πάντως για μας συμπερασματικά αυτό που είναι σημαντικό είναι να μειωθεί ο κίνδυνος δηλαδή τα πλάνα διάσωση θα πρέπει να είναι επί της βάσεως του ότι οι αρχές θα πρέπει μπορούν να τα επιβάλλουν τα πλάνα αυτά όποτε χρειάζεται βάλει. Έχουμε κατεβάσει διάφορες τροπολογίες όπως μια και οι συνάδελφοι. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση και για τα μορατόρια τα είπαμε σε σχέση με την ε, Κεντρική Τράπεζα Είπαμε ότι εμεί δεν θέλουμε να υπάρχουν μορατορία γιατί θεωρούμε ότι αυτό οδηγεί σε άλλα προβλήματα. Δηλαδή αντί να λύνει ε, τα προβλήματα χειροτερεύει τα πράγματα. Τι γίνεται εις βάρος κυρίως των ε, καταθετών, των αποταμιευτών και θα προκύψει μπάνκραν. Δεν έχουμε τις κατάλληλες μεταβλητές παραμέτρους για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. και σε σχέση με τον SSM. Υπάρχουν δηλαδή νομικά ζητήματα. Ή αλλού μπορεί να είναι και θέμα αντιστεγματικότητας Επίσης, έχουμε άλλη τροπολογία για να μην υπάρχει όσον αφορά το μπέλιν αναδρομικότητα. Αναλογικότητα επίσης όσον αφορά τις κεφαλαιοχικές απαιτήσεις όσον αφορά την χρηματοοικονομική δομή της τράπεζας. Υπάρχουν τράπεζες που στέζονται σε καταθέσεις και όχι στις αγορές. Οι συστημικές τράπεζες πάντως να έχουν την υποχρέωση της δημοσιοποίησης των MRL. Πάμε τα βαθιά περίοδο εξαετή και έτσι να συμμορφωθούν οι τράπεζες σε αυτόν τον σημαντικό κανόνα να μην οδηγηθούμε σε προβλήματα στον τραπεζικό τομέα. Και ε, επίσης οι τράπεζες που δεν έχουν εμπειρία από τις αγορές ομολόγων θα πρέπει να συνδυάσουν το MRL με το μετοχικό τους κεφάλαιο. και να δούμε τι θα κάνουμε με το grandfathering σε σχέση με τον οργανισμό CRR. Θα πρέπει να γίνει εναρμόνιση, αλλά χρειάζεται χρόνο. Επίσης, σύμφωνα με τους συναδέλφους, για το buffer των κεφαλικών απαιτήσεων προσοχή στην αυξημένη περιπλοκότητα. Και επίσης, α, είπαμε επίσης για την αναθεώρηση του BRRD. Επίσης, για αυτό το ελάχιστο 8% για τις ε, ζημίες. από πλευράς ομολογιούχων και μετόχων. Εδώ προσοχή να μην θεσπίσουμε κάτι το οποίο να είναι αντισταγματικό σε πολλές χώρες. Α, και κάτι άλλο μας ενδιαφέρει πολύ. Όταν μία τράπεζα μπαίνει σε φάση εκαθάρισης, θα πρέπει να εξετάσουμε το αν μπορεί να γίνει διαρθρωτική μεταρρύθμιση σε αυτήν την τράπεζα, διαρθρωτικές αλλαγές αυτό το σημείο θα πρέπει να προσεχθεί. Βέβαια θα ξανασυναντηθούμε με τον εισηγητή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε περαιτέρω. So we uh, move to the catch the eye and the uh, first speaker is Anne Sander, please. Merci Monsieur le Président.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 να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σχέσεις. Όλη αυτή η συζήτηση για τα MRL πάντοτε είναι πολιτικά φορτισμένη, γιατί το πολιτικό τοπίο είναι κάπως περίεργο. Από τη μία α, οι αριστερές φωνές ισχυρίζονται ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει χώρος για ιδιωτικό banking και ζητάνε περισσότερη πειθαρχία στο τραπεζικό σκηνικό. Δεν είναι όμως συνεπής όταν άκουσα κάποιους συναδέλφους δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με το γεγονός ότι θέλουν πιο ισχυρά πρότυπα αλλά και αναγνώριση των διεθνών προτύπων αντί να υιοθετούμε πιο α, επίοικοι standards. Ίσως θα πρέπει να μιλήσετε λίγο στο τηλέφωνο με τον κύριο Φόξ που ασχολείται με το πακέτο μείωσης των κινδύνων και ζητάει χαμηλότερα πρότυπα στην Ευρώπη σε σχέση με αυτά που ισχύουν διεθνώς. Αυτό που είναι όμως πιο ενδιαφέρον για μένα είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο, στις δύο μεγάλες ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο. Απ' τη μία μεριά έχουμε την πειθαρχία στην αγορά έτσι όπως το θέτει το EPP Με άλλα λόγια, πρέπει ο καθένα να πληρώνει το λογαριασμό που τον αναλογεί, κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύει και για τι τράπεζε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πρότυπα στην Ευρώπη που να εξασφαλίζουν ότι το κράτο δεν θα υποχρεούται να σώσει τι τράπεζε κάθε φορά από μια. Από την άλλη μεριά όμω, οι σοσιαλιστέ εδώ στο Κοινοβούλιο δεν ζητάει τροπολογίες που να ενισχύουν αυτά τα οποία ζητάει η Επιτροπή ή να ενδυναμώνει αυτά που ζητάνε οι αρχές διάσωσης των τραπεζών. Αντιθέτως ζητάνε πιο επική πρότυπα, ζητάνε μεγαλύτερες μεταβατικές περιόδους. Αυτό για μένα είναι απογοητευτικό. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να προσπαθήσει να ακούσει ό,τι φαίνεται να στηρίζει η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και να μην υποκύψει. Με άλλα λόγια να μάθει το μάθημα που μάθαμε από την μη συμμόρφωση με τα πρότυπα σε ό,τι αφορά την κατάρρευση των τραπεζών για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι εδώ κάπως αντιστρέφεται το, το σύνηθες πολιτικό σκηνικό εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τα πακέτα μείωσης των κινδύνων έχουν καταλήξει να είναι άσκηση αύξηση των κινδύνων για κάποιες ομάδες. Πιστεύω θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να πάρω κι εγώ το λόγο, λέει ο πρόεδρος. προτιμώ να λέω αυτά που σκέφτομαι. Και να μην βάζω ταμπέλες στο ένα ή στο άλλο επιχείρημα. Θα ήταν πολύ εύκολο να βρούμε μια απλή γραμμή ερμηνείας σε ό,τι αφορά το τι λέει ο καθένας. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε μια ερμηνεία που να είναι πιο γεωγραφική και λιγότερο πολιτική. Αυτό όμως ήταν λάθος κατά με. Το ουσιαστικό σημείο το οποίο δείχνει να στηρίζει η πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο, που είναι και το πνεύμα της Επιτροπής, είναι το γεγονός ότι πρόκειται για κάτι λογικό. Αλλά και συνεπές με την αρχή του Μπέιλιν. Δεν θέλω τώρα να, να παρεξηγηθώ, αλλά ακριβώς επειδή το bail-in καλύπτει τα πάντα, αυτό είναι ένα διαφορετικό σκεπτικό από τα MRLs. Τα MRLs έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα. Τα δύο αυτά πράγματα λοιπόν είναι διαφορετικά συμπεριλαμβανομένο και το μίνιμουμ 8%. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι σύμφωνα με την Επιτροπή ο εισηγητής προσπάθησε να βρει μια ισορροπία ανάμεσα σε επαρκή ποσά που να μπορούν να εξασφαλίσουν αφενός τη χρηματική σταθερότητα και αφετέρου την διαβίωση των τραπεζών και από την άλλη μεριά τη δημιουργία επαρκών buffers με έναν τρόπο όμως που δεν θα δημιουργεί μη σταθερότητα. Ο προσωπικός μου ορισμός, σε αφορά τη μείωση των κινδύνων, είναι να προσπαθείς να μην δημιουργείς καταστάσεις που προκαλούν κινδύνους. Ή το μορατόριο, για παράδειγμα, που συζητήσαμε. Δεν μπορούμε να ονομάσουμε το μέτρο αυτό μέτρο μείωσης κινδύνου. Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο σε ό,τι αφορά τα τίλαξ, τη συνολική ικανότητα απορρόφηση ζημιών, σε ό,τι αφορά τις πιο πολύπλοκες και δύσκολες να διασωθούν τράπεζες, το βρισκολογικό να είναι ένα σημείο αναφοράς το τιλάξ Ένα εργαλείο που μπορεί να απλοποιήσει και να βοηθήσει στη διάσωση των τραπεζών. Αν έχεις Μία τράπεζα που πρέπει να διασωθεί και μία τράπεζα που πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί και πάλι έχει δύο διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι διαφορέ. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευχέρεια των αρχών, βεβαίω και θα πρέπει να είναι στην ευχέρειά του το εκάστοτε σχέδιο δράση. Σε ό,τι αφορά να αποφασίσουν κατά πόσο θα πρέπει να διασωθεί μια τράπεζα ή όχι. Αυτό που κάνουμε όμως εμείς όταν νομοθετούμε είναι να θέτουμε ένα πλαίσιο, να πλαισιώνουμε την αρχή αυτή και να λέμε πού μπορεί να είναι ευέλικτη, ποιες είναι οι ευθύνε που θα πρέπει να έχει εκάστοτε αρχή και ποια είναι και τα πρότυπα που θέτουμε. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας διαφορετικά. Ποιο το νόημα του να θεσπίζουμε κανονισμούς πρώτο, δεύτερο κτλ μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων για να καταλήγουμε στο ότι είναι στην ευχέρεια του εποπτικού μηχανισμού. Όχι. Νομοθετούμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και θέτουμε και το όριο μέχρι πού φτάνει η ευχέρεια της κάθε εποπτικής αρχής. Θεωρώ ότι να πλαισιώνουμε λοιπόν την ευχέρεια και την ευελιξία της κάθε εποπτικής αρχής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε. Όχι βεβαίως ενάντια, δεν μπορούμε να δένουμε τα χέρια της εποπτικής αρχής. Θα πρέπει όμως να θέτουμε τα όρια μέσα στα οποία θα μπορεί να κινείται η κάθε εποπτική αρχή, αρχή διάσωσης κτλ και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στην κατάσταση του κάθε τραπεζικού ιδρύματος. Θεωρώ λοιπόν ότι αν κρατήσουμε την ιδεολογία έξω από τη συζήτηση αυτή και συζητήσουμε με ένα ρεαλιστικό τρόπο, παίρνοντας, λαμβάνοντας υπόψη μας αυτές τις αρχές τις οποίες ε, ε, στήριξε και ο εισηγητής, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν ε, άλλοι που θέλουν να μιλήσουν. Όχι, το λόγο έχει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τον Σβέν Γκίγκολτ για την γενικότερη κρίση του, για το εάν έχουμε τις σωστές απόψεις και ποιες απόψεις ε, πρέπει να έχουμε. Νομίζω, ε, εντάξει, καλά τα πήγα, ε, κάνα 8 ή 9 στα 10 φαντάζομαι. Ε, και τέλος πάντων μοιάζει με στήριξη ούτως ή άλλως. Γενικότερα νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ένα πράγμα. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση ή ιδέα που έχει σχέση με τις μελλοντικές διαδικασίες που θα αποδυναμώσει την οδηγία. Έχει αλλάξει το τοπίο πάρα πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια με όλες αυτές τις διαφορετικές νομοθεσίες, ειδικά για τις τράπεζες, με τις οδηγίες κεφαλαϊκής επάρκειας και την PRD. Ε, θα ήθελα εγώ να επισημάνω ένα πράγμα που έχει κρίσιμη σημασία για την οδηγία διάσωσης ε, των ε, τραπεζών, η οποία πλέον περνάει στην πραγματικότητα. και βεβαίως ε, η πειθαρχία των αγορών εξαρτάται από το ότι τα πάντα υπόκεινται σε bail-in. Αλλιώς ε, ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ναι. Κάποιες ειδικέ δόσεις του κεφαλαίου που υποτίθεται ότι υπόκεινται στο bail και θα τιμολογηθούν ανάλογα, αλλά ε, μετά δεν θα υπάρχει πίεση στις τράπεζες, στις χρηματαγορές. Γι' αυτό ήμουν ε, αυστηρός όσον αφορά το λέξει στην πρόταση μου, γιατί εάν ξαφνικά επεκτείνουμε το ε, χρέος αυτό μιας συγκεκριμένη ε, κατηγορία, θα το θεωρήσουν οι τράπεζες ότι αυτό υπόκειται σε Μπέιλιν να το επαναλάβω, η πειθαρχία των αγορών είναι ακριβώς ε, μία από τις ε, σημαντικότερες ε, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς πίεσης. Γιατί οι τράπεζες δεν είναι απομονωμένες. Πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούν την οικονομία. Αλλιώς η οικονομία θα μαραζώσει. Οπότε όταν αναπτύσσεται η οικονομία οι τράπεζες είναι και πιο σταθερές ε, και το αντίθετο ανεξαρτήτως νομοθεσίας. Όσον αφορά λοιπόν την οδηγία BRD έχουμε πρώτα απ' όλα την σειρά του Μπέιλιν και άλλα μέσα ε, για τράπεζες οι οποίες χρεοκοπούν αλλά έχουμε και τα σχέδια διάσωση που επισήμανε ο κύριος Φουρτασούν και θεωρώ ότι στι μελλοντικέ διαδικασίε πρέπει να είμαστε σαφής ε, απέναντι στις ε, αρχές διάσωσης ότι πρέπει να υπάρχουν ε, σχέδια τέτοια, όχι ενδεικτικά μέτρα. Καμιά φορά όταν ακούω τέτοιες αρχές θέλουν περαιτέρω κατεύθυνση τους, έχω δεν έχετε συντάξει τέτοια σχέδια με την ιεραρχία. Συνολικά λοιπόν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το που βρισκόμαστε σήμερα με το που βρισκόμασταν πριν από μερικά χρόνια. Και τώρα έχουμε επίσης το τηλεκτόπιο το οποίο παρέχει περισσότερη σταθερότητα. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση στη δική μου την έκθεση ότι ο περιορισμός του θα πρέπει να είναι περιορισμός του MRL. Πρέπει να το θυμάμαστε αυτό. Και αυτό υπάρχει επίσης ε, και στην σκέψη μου ότι τα πάντα πρέπει να υπόκεινται σε Μπέιλιν. Ελπίζω λοιπόν να κάνουμε μια κοινή ε, προσπάθεια. Πολλοί μίλησαν για το ότι πρέπει να έχουμε εξαιρέσει και υπάρχουν και σχετικέ τροπολογίες. Όλοι ήθελαν επίση ε, εξαιρέσει από την οδηγία BRD. Ε, θα είναι μετά σαν ελβετικό τυρί γεμάτο τρύπε. Και δεν είναι σωστό και αυτό. Οι τράπεζες ε, πρέπει να θεωρούνται ως ιδρύματα με κινδύνους. Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχουν κάποια ειδικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα λάβουμε υπόψη, αλλά θα ήθελα να είμαστε πολύ περιοριστικοί όσον αφορά τις εξαιρέσεις. Αλλιώς μετά δημιουργούμε αυτό το οποίο είπα το ελβετικό τύρι. Για την κατεύθυνση τώρα που θα δίνεται. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και για το μορατόριο επίσης, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πηγαίνουμε μάλλον προς την κατεύθυνση την οποία πρότεινα. Ίσως ε, θα έπρεπε να, κάνουμε, να διευκρινίσουμε υπό ποιες συνθήκες μπορεί να υπάρξει ένα συντομότερο μορατόριο και να είμαστε ρεαλιστές και να επιτύχουμε κάτι. Σας άφησα όλους, ε, σημείωσα με καλή διάθεση και νομίζω ότι με την αξιολόγηση του Sven Giggold καλά τα πήγαμε. Σας ευχαριστώ. Και όπως είπατε καλό είναι να έχουμε καλή διάθεση. Λοιπόν. Η επόμενη προθεσμία είναι η ψηφοφορία 16-17 Μαΐου. Έχουμε λοιπόν χρόνο μπροστά μας για να εργαστούμε προσεκτικά. για να προετοιμάσουμε τις συμβαστικές προτάσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση ως αποτέλεσμα της ε, έκθεσής σας για να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο ήδη τον Μάιο-Ιούνιο για να ολοκληρωθεί ρεαλιστικά αυτή η νομοθεσία πριν το τέλος του έτους. Ένα θεμελιώδες κόμμα. Το χειρότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, αν είναι να ολοκληρωθεί το τραπεζικό πακέτο και να εισαχθούν τέτοια μέτρα μείωση του κινδύνου όπως το MRL είναι να μην τελειώσουμε εγκαίρω. Οπότε ε, πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν την έκθεση, ακολουθούν τροπολογίες ε, και βλέπουμε ήδη την δυνατότητα συμβιβασμών. Θα έλεγα λοιπόν ότι μετά το την ε, σημερινή ημέρα. Είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα αυτό και σας καλώ να το σεβαστείτε όλοι για να κάνουμε την... το καθήκον μας ως νομοθέτες και να μπορέσουμε να καταλήξουμε έγκαιρος. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, Πέτερ Σίμων και πάλι πολλές τροπολογίες αναμενόμενο όμως Α, λογικό για μια τέτοια έκθεση ε, δεν είναι και εύκολο βεβαίω, δεν είναι και εύκολο δουλειά σου Πίτερ νομίζω ότι μπορείς Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την εμπιστοσύνη του Προέδρου ε, για το ότι μπορώ να αντιμετωπίσω 1300 ε, τροπολογίες ε, που υποβλήθηκαν. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι οι συνάδελφοι τα υπέβαλαν όλα αυτά. Βεβαίω πράγματι αν σκεφτούμε την περίοδο 2009-2014 είχαμε εκθέσει με 2.500 τροπολογίες οπότε πάλι φτύνα την γλίτωσα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διαβάσω την κάθε τροπολογία οπότε είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση και αν τα καταφέρουμε νομίζω να πάμε κάποια στιγμή τον Μάιο στην ψυχοφορία θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ και βεβαίως υπάρχει και το Πάσχα στη μέση δύσκολα. Λοιπόν, να έρθουμε στα βασικά σημεία που αναφέρονται στις ε, τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στην ε, επανεξέταση του Trading Book. Κάποιες ε, τροπολογίες μιλάνε για το να αφήσουμε το όριο των ιδιών κεφαλαίων στο 65% των απαιτήσεων της Βασιλείας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκάθαρα ζήτησε μια σταδιακή προσέγγιση και εγώ θεωρώ ότι η πρότασή μου χρειάζεται μια πενταετή μεταβατική περίοδο. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας καλός συμβασμός, αλλά είναι συζητήσιμο. Επιπλέον η φάση της εφαρμογής ε, που ε, θα εκτείνεται σε τρία χρόνια θα μας δώσει και θα δώσει την Κομισιόν επαρκή χρόνο για να αντιδράσει στην Βασιλεία. Μετά, δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης όσον αφορά τα ρέπος στο πλαίσιο του δίκτυου ρευστότητα και την λεγόμενη ασυμμετρία στην αντιμετώπιση αυτών. Εδώ πέρα η Κομισιόν αποφάσισε εσκεμένα να αποκλίνει από τα της Βασιλείας ε, για να αποδυναμωθεί αυτή η ασυμμετρία. Η πρότασή μου είναι η ασυμμετρία αυτή να αυξηθεί με το να μπορούμε να αντισταθμίσουμε τα repos με τα reverse repos όπως λέγονται για να σταθεροποιηθεί η σχετική αγορά. Πολλοί συνάδελφοι έχουν υποβάλει εδώ πέρα τροπολογίες για να διαγραφεί τελείως η ασυμμετρία στην αντιμετώπιση τους πράγματα τα οποία γνωρίζουμε από το NSFR. Γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω πως η ασυμμετρία στην αντιμετώπιση είναι κάτι το οποίο θέλαμε ρητά. Δεν είναι κάποιο συντακτικό λάθος και αυτή η ρύθμιση έγινε ηθελημένα. Και η Ευρωπαϊκή ε, Τραπεζική Αρχή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρούν ότι πρέπει να μείνουμε στη, στα της ε, Βασιλείας. Ε, προσωπικά λοιπόν έχω βάλει και κάποιες ε, τροπολογίες και είμαι αρκετά επιφυλακτικός για αυτό το οποίο λέει η Κομισιό να πάμε πέρα από την Βασιλεία, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει εδώ πέρα μια συζήτηση εις βάθος. Τίλεκ, το τρίτο απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν και το πώς θα εφαρμοστεί για την δεσμευτικότητα της σχετικής ρήτρας. Κάποιοι συνάδελφοι επίσης πρότειναν για συστημικά ιδρύματα να υπάρξουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσει που κυμαίνονται από το 8% μέχρι 13,5% σε άλλες, συνα... σε άλλες προτάσεις συναδέλφων για το ποσοστό χρέους ε, θεωρώ ότι αποφασιστικό ρόλο θα παίξει το εάν υπάρχουν τράπεζες συστημικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα έχουμε διαφορετικές απαιτήσεις που κυμαίνονται από το 10% μέχρι το 6% μέχρι αυτό το οποίο αποφασίστηκε στην ε, Βασιλεία τον Δεκέμβριο για 50% του κεφαλαιακού αποθεματικού. Έχουμε λοιπόν πολλές συζητήσεις στις επόμενες εβδομάδες, αλλά θα ήθελα να πω ότι η δική μου η προσέγγιση να μείνουμε στο 4% για ιδρύματα τα οποία έχουν παγκόσμια συστημική σημασία είναι νομίζω μια ισορροπημένη προσέγγιση γιατί ευρωπαϊκές ε, τράπεζες με παγκόσμια συστημική σημασία ήδη εκπληρώνουν ε, και με το παραπάνω σήμερα αυτήν την απέτηση. Αν λοιπόν ανέβουμε παραπάνω και κινηθούμε ε, εκεί όπου βρισκόμαστε περίπου σήμερα, νομίζω αντικατοπτρίζουμε την σημερινή τραπεζική πραγματικότητα ως έχει και αφενός αποφεύγουμε την υπερβολική επιβάρυνση αλλά από την άλλη έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο μόχλευσης από αυτό το οποίο μας πρότεινε η Κομισιόν. Λίγα λόγια για τις IPU, ένα άλλο σημαντικό θέμα στις ε, τροπολογίες έχουμε το θέμα δηλαδή του ποιες συστημικές τράπεζες οι οποίες ε, δεν έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ακριβώς να υποχρεωθούν να ιδρύσουν μια άλλη επιχείρηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα υπόκειται σε εποπτεία. Εδώ πέρα ε, λοιπόν οι συζητήσει είναι το εάν και τι μορφή θα πρέπει να ε, έχει μια τέτοια IPU. Δεν θέλω τώρα να προδικάσω εγώ την συζήτηση αλλά να γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι θέλουν να γίνει συζήτηση. Κάτι άλλο το οποίο παίζει βασικό ρόλο στην έκθεσή μου και θα ήθελα εδώ πέρα να κλείσω την ε, σύντομη εισαγωγή μου κάτι το οποίο οδήγησε επίσης σε πολλές προτάσεις είναι η λεγόμενη αναλογικότητα χάρηκα ε, για το ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτό και έκαναν πολλές προτάσεις. Ο συνάδελφος των Πρασίνων εδώ πέρα αφενός οι Πράσινοι έκαναν πολλές προτάσεις για ελάφρυνση των μικρών ε, και μη περιπλοκών τραπεζών όπως και ο συνάδελφος εδώ από το Τσεσού επίσης έκανε την ίδια πρόταση αλλά επίσης ε, θα πρέπει, λένε, να συνδέονται αυτά με υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τέτοια τραπεζικά ιδρύματα που έχουν ένα λόγο ιδίου κεφαλαίου 15% και ένα ποσοστό χρέωσης 6% για να μπορέσουν να ωφεληθούν. Δηλαδή από τη μία ελαφρύνσης αλλά ως αντάλλαγμα από την άλλη αυξημένες απαιτήσει για όσους θα έχουν αυτήν την ελάφρυνση. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση που οπωσδήποτε θα την συζητήσουμε. Άλλες τροπολογίες ζητάνε ε, να αυξηθεί το κατόφλι γιατί λένε τι είναι μικρό, 1,5 δισεκατομμύριο σε μια χώρα όπως η Μάλτα ε, είναι ήδη πάρα πολλά σε μια χώρα όπως η Γερμανία με το ανάλογο ΑΕΠ είναι κάτι το μικροσκοπικό. Οπότε θα πρέπει ακριβώς να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη λύση. Οπωσδήποτε κατατέθηκαν εδώ πέρα τροπολογίες και τροπολογίες οι οποίες πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση του περιορισμού τέτοιων τραπεζών οι οποίες εξαιρούνται λόγω του μεγέθους τους ε, και να περιοριζόμαστε σε τράπεζες που έχουν ένα 10% της αγοράς στην χώρα τους. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε χίλιες τράπεζες σε μια χώρα και 900 από αυτές είναι μικρές, παρόλα αυτά ε, το πολύ 100 από τις 900 θα πρέπει να εξερευθούν και οι 800 παρά το ότι είναι εξίσου μικρές θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως CRRD και τα λοιπά και όχι στην πλήρη έκταση όπως δηλαδή είχε προτείνει η Κομισιόν και εγώ με μια πιο ελαφριά μορφή. Εδώ πέρα θα οδηγηθούμε σε προβλήματα σε χώρες όπου υπάρχει μία μικρή συγκέντρωση της αγοράς και δεν νομίζω άλλωστε ότι είναι η δουλειά μας εδώ πέρα να νομοθετήσουμε ανάλογα με το ερώτημα εάν προτιμούμε αγορές πιο, με πιο μεγάλη συγκέντρωση ή με πιο ε, μικρή συγκέντρωση. Πρέπει να δούμε τα ιδρύματα, της ε, τράπεζες και από εκεί να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την επικοδομητική συνεργασία. Αναμένω και τις συζητήσεις που θα έχουμε, τις συναντήσεις, την ανταλλαγή απόψεων με τον συνάδελφο Χέκμαρκ για να καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα το οποίο θα κάνει πιο σίγουρες τις τράπεζες και θα είναι και κοντά στην σημερινή πραγματικότητα. Μέχρι τον Μάιο λοιπόν, αν γίνεται, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας για να μπορέσουμε να πάμε μέχρι το Μαΐο στην Ολομέλεια και ίσως τον Ιούνιο να πάμε στις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Αν το καταφέρουμε αυτό, έχουμε μια ελπίδα να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος φέτος, κάτι το οποίο έχει την σημασία του είναι πράγματα που ε, θα πρέπει να τεθούν ενισχύ από το 2019. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Thank you. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω, ε, ε, δεν μπορώ να, να μην πω στον πειρασμό να αναρωτηθώ ότι οι πολιτικοί μας έχουν την ίδια τροπολογία αναλογικότητα και πράσινη. Τέλος πάντων. Πρέπει, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι επιλογή, υποχρέωση είναι. Ο Μαρκάρας είναι ο πρώτος πληστής του λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πέτερ, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που ακούω ότι θέλετε να ολοκληρώσετε το θέμα φέτος Βεβαίως η προεργασία που γίνεται με τους γεωδησίτες νομίζω θα μας βοηθήσει. Εξαρτήτως του τι θα γίνει με τις τροπολογίες είμαστε σε καλό δρόμο. Ε, σοβαρά προβλήματα έχουμε λίγα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τον στόχο της όλης διαδικασίας. Δεν ναι, θα ήθελα λοιπόν να τα επαναλάβω όλα για την αναλογικότητα και τον ορισμό θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε το κατόφλι των 500 εκατομμυρίων ευρώ για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Συμφωνούμε για τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων. Επίσης για το ερώτημα τώρα θα ήθελα να πω ότι είναι καλό να λάβουν υπόψη αυτά τα οποία είπε η τελευταία έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το ESRB. Για τις παγκόσμιες ε, προδιαγραφές ε, ε, για την ομάδα μου είναι σαφές ότι πρέπει να πάμε στην απέτηση του 3% για το αποθεματικό για τις παγκόσμια σημαντικές συστημικές τράπεζες θεωρούμε να υπάρξει μια ρύθμιση της εφαρμογής της βασιλείας για τις συστημικές τράπεζες το απορρίπτουμε γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί κάτι το επιπλέον σε σχέση με τις απαιτήσει της βασιλείας για το NSFR και το διαρθρωτικό ποσοστό ρευστότητας θα πρέπει να συμμορφωθούμε με τη Βασιλεία και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε το 5% όσον αφορά τώρα τις αλλαγές στην ασύμετρη μεταχείριση των ρέπος και reverse ρέπος. Ναι, είμαστε υπέρ για αποφάσεις επίπεδου 1 και κατά μιας πράξης κάτω εξουσιοδότηση ή αυτόματης προσαρμογής για το ερώτημα των ε, trading books είμαστε πάρα πολύ κοντά και έχουμε μια προθεσμία τουλάχιστον τριών ετών για το ζήτημα ε, ψηφιακά και επενδύσεις σε λογισμικό συμφωνώ με αυτό το οποίο λένε σχεδόν όλες οι ομάδες δηλαδή θα πρέπει να εξετάσει το θέμα Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για τις επενδύσεις ε, ιδίων μέσων σε λογισμικό. Έχουμε τώρα το άρθρο 113 της Οδηγίας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια για τα τραπεζικά ιδρύματα με ένα προφίλ κινδύνου. Επίσης, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τακτική εξέταση της μακροπροληπτικής τάσης για το θέμα του ΤΙΛΑΚ. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς τις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες σε τρίτες χώρες τις αρχές ε, διασύσου θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να φέρουν τις δικές τους προδιαγραφές σε σχέση με τις παγκοσμίες και το 75% αυτών που έχω προβλήματα στο θέμα της αποζημίωσης κατά την απόψή μου χρειάζεται λιγότερη εθνική διακριτική ευχέρεια αλλά πιο ευέλικτος ευρωπαϊκός κανονισμός όσον αφορά το κατόφλι για την δε δημοσίευση των ποσοστών αποζημίωσης είναι κάτι το οποίο απορρίπτουμε. Για τον δε κίνδυνο του κάθε τραπεζικού ιδρύματος το βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι ακριβώς ο κίνδυνος για δεν πράσινο ή κοινωνικό συντελεστή επιχειρηματικότητας χρειαζόμαστε νομίζω περισσότερα στοιχεία και σοβαρότερη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Οπότε θα πρέπει να δούμε και την σχέση αυτού του κανονισμού με την πρόταση της Κομισιόν του Μαρτίου και να αποφευχθεί η σύγχυση. Τέλος, για το θέμα αποκάλυψης κλιματικών κινδύνων προτείνω να εξετάσουμε πρώτα απ' όλα αν η εισαγωγή μιας τέτοιας κατηγορίας κινδύνου δικαιολογείται και αν ναι πώς θα πρέπει να οριστεί. Θεωρώ ότι θα πρέπει ακριβώ να δούμε το τι γίνεται γιατί έχουμε ε, διαφορετικές απαιτήσεις. Το ένα είναι απάντηση στην Βασιλεία και το άλλο είναι μια επιπρόσθετη απέτηση. Ναι, εφαρμογή αυτή τη στιγμή όμως όχι. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση. Thank you. Και εμείς ευχαριστούμε, λέει κύριος Γκουαλτιέρ γιατί το λόγο στον κύριο Φως. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους χιοδησηγητές αλλά και τον εισηγητή για τη γραμματεία γιατί ε, διεκπαιρέωσαν ε, όσο πιο μπορούσαν τις τροπολογίες για να είμαστε στο χρόνο διαγραμμόπουσαμε και πριν δεν καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οι διεθνείς τράπεζες που έχουν πολλές θεατρικές θα πρέπει να έχουν ένα IPU ή αν έχουν ε, σύνδεγιο 30 δις. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ και κοιτώντα τι τροπολογίε βλέπω ότι και άλλοι συναδελφοί πρεσβεύουν τα ίδια και συμφωνώ με τι τροπολογίε που λένε ότι αυτό θα πρέπει να απαλληφθεί τελείω. Εάν ε, χρειάζεται ένα IPU, τότε νομίζω ότι χρειάζεται ένα κατόφλι 50 δι και άρα χρειάζεται να έχουμε δύο IPU. Και έτσι θα κάνουμε τα ίδια με του Αμερικανού και δεν θα έχουμε τίποτα αρνητικέ συνέπειε από άλλε αγορέ τώρα Όσον αφορά το net stable ratio, πιστεύουμε ότι τα παθητικό που σχέση με παράγωγα θα πρέπει να το προσέξουμε να δούμε αν είναι πραγματικό και γνήσιο. Να δούμε μπορεί να συμβαστούμε. Κάποιοι συναδελφοί επίσης δεν θέλουν να υπάρχει σταθερό προαπαιτούμενο χρηματοδότησης. Αυτό είναι υποτίμηση του κινδύνου. Τώρα όσον αφορά το ρευστό προς αντιστάθμιση η αμοιβή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν αναλογική προσέγγιση για τις μικρές και απλές τράπεζες. Δεν σύμφωνα ότι θα πρέπει να έχουμε ένα pay ratio σαν ανώριο για την μέση αμοιβή υπαλλήλου. Είπαμε να επαναφέρουμε το 103 σύμφωνα με το CRD. για κεφαλαιογικά και μη μέτρα όσον αφορά τον κίνδυνο. Και αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις τράπεζες. Επίσης το ίδιο όσον αφορά τον λόγο μόχλευσης σύμφωνα με τη Συμφωνία της Βασιλείας και από αυτόν τον λόγο να εξαιρεθούν τα αποθεματικά των τραπεζών. Και όπως και στην αδελφή του S&D, Άλντε και ΕΛΚ και εγώ έχω κάποιες τροπολογίες όσον αφορά τους aggregators της αγοράς ούτως ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τιμές όλη της αγοράς οι τραπέζες να είναι ξεκάθαρο το τοπίο και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές υπηρεσίες οι τράπεζες διάφοροι συναδελφοί υπέβαλαν τροπολογίες τόσο ώστε κάποιο λογισμικό να εξαιρείται από τα στοιχεία του ενεργητικού όμως αυτό είναι αντικίνητρο για επενδύσεις όσον αφορά το green scaling factor και τα κίνητρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε αυτή τη δέσμη μέτρων να υπάρχει τέτοιου είδους κύρωση. Ούτε συμφωνώ να είναι 0% ο υπολογισμός του δημοσίου χρέους. Και χαίρομαι που και να πιστεύουν το ίδιο. Σβέν Γίγκολ, θέλω να σε γλώσσα το ECR δεν θέλει να απονευρώσει τα πρότυπα της Βασιλείας. Θέλουμε η νομοθεσία μας να είναι ρεαλιστική. Δεν θέλουμε φτιασίδια πράσινα και οικολογικά που θα δυσκολέψουν τις συναλλαγές. Και θα συνεργαστούμε, ελπίζω, με τον εισηγητή και τους κοιόδους εισηγητές. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το ποια θα είναι τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον έχει να κάνει με το ποια θα είναι τα πρότυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που αποφασίσετε να φύγετε, λέει ο Πρόεδρος. Βεβαίως όμως και <clears throat> καταλαβαίνω η κυρία Νατ Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θέλω να κάνω κάποια γενικά σχόλια αρχικά πριν επισέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες κάποιων τροπολογιών. Θέλω να τονίσω ότι ο βασικός μου στόχος είναι να ευθυγραμμιστούμε με τα διεθνή πρότυπα την αύξηση της σταθερότητας αλλά και επιπλέον μείωση των κινδύνων είναι πολύ σημαντικά σημεία σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Βεβαίως και έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Όπως είπα, είμαι υπέρ της ευθυγράμμισης με τα διεθνή πρότυπα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν δεν μπορώ να στηρίξω προτάσεις που έκαναν κάποιοι συνάδελφοι που θα μπορούσαν ίσως να καταλήξουν σε ξεχωριστά ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τη μείωση των ρίσκων στον χρηματοοικονομικό τομέα. Πρέπει να κάνουμε πρόοδο όπως ξεκινήσαμε στην Βασίλεια. Θέλω να τονίσω κάποιες από τις προτεραιότητές μου Πρώτα απ' όλα, σε τη φορά το CID, χαίρομαι που βλέπω ότι μια ευρεία πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο. Θεωρεί ότι προκειμένου να εφαρμοστούν α, τα πρότυπα που θέλουμε θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό σε 40 δισεκατομμύρια. Επιπλέον συμφωνώ, θεωρώ ότι είναι αρκετή μεταβατική περίοδος των τριών ετών. Δεύτερον, πολλοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τεχνικά προβλήματα, κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνη. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τα MRLs, και τις τροπολογίες και πάλι πιστεύω στην ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα ο συντονισμός αυτός θα εξασφαλίσει περισσότερο την ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να δημιουργεί επιπλέον κινδύνους. Ένα τέταρτο σημείο το οποίο έθιξα ήδη τον Δεκέμβριο συμφωνώ με τον εισηγητή ό,τι αφορά ε, το ότι πρώτα θα πρέπει να είναι πιο προσαρμόσιμη σε, για μικρότερες τράπεζες. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία για το σημείο αυτό, για τράπεζες δηλαδή, οι οποίε θα πρέπει να, είναι, ε, να υπόκειται σε ένα διαφορετικό καθεστώ. Θεωρώ ότι στόχος της συζήτησης αυτής είναι να είμαστε πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, προνοητικότητα χωρίς να υπερεκτιμούμε τους κινδύνους. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις δημόσιες τράπεζες. Εδώ προτείνουμε μία τροπολογία για να περιοριστούν οι εξαιρέσεις μόνο στις εθνικές τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε κυβερνήσεις αλλά και σε οργανισμούς που προσφέρουν δημοσίες υπηρεσίες. Όπως έθιξα και τον Δεκέμβριο, αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Προτείνω την τροπολογία του εισηγητή και πιστεύω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμούς. Τέλος και το πιο ευαίσθητο σημείο για μένα Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τις ανακεφαλοποίησεις, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό συμβασμό μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μπροστά μας μήνες από, για διαβουλεύσεις, αρκετά ζητήματα θα συζητηθούν. Ανυπομονώ για μια αγαστή συνεργασία Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα πετύχουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Μάιο. Ο κύριος Μακάρτη έχει το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες να εισάγουμε μεγαλύτερη αναλογικότητα, θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό και με μια διαφορετική οπτική γωνία θα πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία σε ό,τι αφορά τι μικρότερες τράπεζες. Όμως το σύνολο του πακέτου αυτού θα πρέπει να επικεντρωθεί στα πιστοτικά ιδρύματα χωρίς να συμβιβαζόμαστε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς για τις τράπεζες. Προτείνουμε λοιπόν τροπολογίε σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Σε ό,τι αφορά το 5% που προτείνεται από τον όσα θεωρούμε ότι είναι πιο επικοδομητικό από το 3%. Ο δείκτης μόχλευσης που προτείνουμε εμείς θα πρέπει να είναι αναλογικός με το εκάστοτε επενδυτικό ίδρυμα να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6% για συγκεκριμένα ιδρύματα και για όλα τα υπόλοιπα να βρίσκεται στο 3%. 100. Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό τώρα του μηχανισμού μόχλευσης, δεν θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να υπάρχουν παρεκκλήσεις από τα διεθνή πρότυπα. Το ίδιο ισχύει και για το TILAC που θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως χωρίς παρεκκλήσεις. θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο απόθεμα που δεθέτουμε μπορεί να μην είναι αρκετό για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικέ τραπεζικές κρίσεις, άρα θα πρέπει ίσω το τίλακ να αυξηθεί. Ανάλογα μέτρα θα πρέπει να εισαχθούν σε εθνικό επίπεδο και για συστημικές τράπεζες. Προτείνουμε λοιπόν στην τροπολογία μας για το άρθρο 92A να αυξηθούν σταδιακά τα αποθεματικά. Σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα, θεωρούμε ότι όλες οι υποχρεώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη νομική επιτυχία συμφωνούμε με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύει αναλογικότητα ανάλογα με την τράπεζα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις υποδομές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύσουν ούτως ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν τράπεζες με μικρότερα κεφάλαια. Θεωρούμε ότι αυτό δεν θα αποδυναμώσει τις εποπτικές αρχές, οι οποίες και θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις άμεσα όταν θεωρούν ότι υπάρχει επικείμενος κίνδυνος. Επιπλέον, δεν επιθυμούμε τη διαγραφή του άρθρου 103 και έχουμε ιδιαίτερες ανησυχίες και δεν θεωρούμε σκόπιμες τις α, εξαιρέσεις δεν συμφωνούμε τέλος με την Επιτροπή. Θεωρούμε ότι κάποια ζητήματα που θίγονται στις τροπολογίες μας θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον ε, δημιουργία πλαισίου και βεβαίως προσβλέπουμε σε μια αγαστή συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τους πράσινους, ο Σβέν. Θέλω απλώς να σας πω ποιες είναι οι δικές μας γενικές γραμμές. Υπάρχουν τόσες πολλές λεπτομέρειες που θα πρέπει να θίξουμε στις διαπραγματεύσεις. Θεωρούμε όμως ότι το κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να σκεφτεί λίγο περισσότερο την Τραπεζική Ένωση και τη συζήτηση που αυτό δημιουργεί. Από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε την φιλοδεξία να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση. Υπάρχουν όμως ανησυχίες ότι αν υπάρξει μια τοπική κρίση η έλλειψη ενός γενικότερου ευρωπαϊκού αποθεματικού θέτει σε κίνδυνο αυτή την τραπεζική ένωση και μπορεί και να οδηγήσει σε διαφυγή κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε και ζητήματα αξιοπιστίας ό,τι αφορά τις αρχές διάσωσης. Είναι ανάγκη λοιπόν να, έχουμε, να ενδυναμώσουμε τον διαμοιρασμό του κινδύνου και ούτως ώστε αυτό να είναι πολιτικά αποδεκτό θα πρέπει, να, θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι στρατηγικές μείωση των κινδύνων. Θέλουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, άρα ως Κοινοβούλιο είναι ανάγκη να αναλάβουμε ηγετική θέση ε, σε ό,τι αφορά την μείωση των κινδύνων, χωρίς παράλληλα να εμποδίζουμε τις πρόοδους στο Συμβούλιο. χωρίς να ευθυγραμμιζόμαστε με αυτούς που δεν επιθυμούν την από κοινού ανάληψη των ευθυνών για τους κινδύνους. Ο εισηγητής πιστεύουμε σε ό,τι αφορά το σκεπτικό του έχει μια παρόμοια γραμμή και αυτό μας, κάνει, μας χαροποιεί. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να εξετάσουμε και τις λεπτομέρειες υπάρχουν ήδη τράπεζες οι οποίες υπό την ε, διεθνή οι οποίες ε, έχουν ε, χαμηλά αποθεματικά. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι κανόνες που έχουμε εφαρμόσει μετά την κρίση έχουν οδηγήσει σε πολύ πολύπλοκους κανόνες ό,τι αφορά συστήματα αναφοράς. Ευχαριστούμε και πάλι τον εισηγητή. Δεν είμαστε υπέρ του να έχουμε ένα χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τις μικρές τράπεζες. Θέλουμε να υπάρχουν πιο απλοποιημένοι δείκτες μόχλευσης σε ό,τι αφορά τις μικρότερες τράπεζες και να, να απλοποιηθούν και όλα αυτά τα συστήματα αναφοράς για τις μικρότερες τράπεζες. Σε ό,τι αφορά και το σχόλιο του εισηγητή μεταξύ των πρασίνων στην Ευρώπη και ενός τοπικού κόμματος, η συμφωνία αυτή, η συμμαχία αυτή υπάρχει, γιατί βεβαίως είμαστε πιο κοντά σε αυτές τις μικρές τράπεζες. Το feedback που έχουμε είναι ότι είναι σε θέση να έχουν, να ανταποκριθούν σε πιο ψηλά, στις ανάγκες πιο ψηλής, υψηλής κεφαλαιοποίησης χωρίς όμως να τις επιβαρύνουμε με δεκάδες απαιτήσει αναφορών. Η Γερμανία έχει ακόμη πολλές μικρές τράπεζες, κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Ακούμε όμως τα ίδια παράπονα από πιστοτικά ιδρύματα και από τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει όλο αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Δεν θέλουμε να βγάλουμε από την αγορά τα μικρότερα ιδρύματα. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο δραστική ατζέντα να σηκώσουμε το βάρος αυτών των πολύπλοκων κανονισμών ενώ παράλληλα να προστατέψουμε τις φιλοδοξίες του πακέτου αυτού. Κύριε Φόξ, επειδή συζητήσατε με τον κύριο Καμάλ, βεβαίως καλωσορίζουμε ε, το ότι συμμορφώνεστε με τα διεθνή πρότυπα. Σε ό,τι όμως αφορά την καθαρή σταθερή χρηματοδότηση, θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Θεωρώ ότι θα πρέπει από κοινού να υπερασπιστούμε αυτά τα διεθνή πρότυπα, όχι να τα αποδυναμώσουμε όπως προτείνεται σε κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι τροπολογίες μας αποσκοπούν κατά κάποιο τρόπο να καλύψουν την δυνατότητα να μπορεί να διορθωθεί μέσω της πραγματικής οικονομίας ότι αυστηρό μπαίνει σαν κορσέ στις τράπεζες για τα δάνεια προς τις ΜΜΕ και προς νοικοκυριά. Αναζητείτε επομένως πιθανότητα λύσεις να ενθαρρύνουμε κάποιες πρακτικές, να αποθαρρύνουμε άλλες. όπως ακριβώς και το τραπεζικό πακέτο επιδιώκει. Θα δούμε τι θα γίνει με τα κατόφλια, με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τις επενδύσεις σε πρασίνη ενέργεια, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι σημαντικό παράλληλα να υπάρχουν κυρώσεις για επενδύσεις που οδηγούν σε εντατικότερη χρήση άνθρακα. Αυτά που λέει η Επιτροπή μας οδηγούν σε κάποιες επιφυλάξεις να έχουμε βιωσιμότητα από πλευρά συνεργειακής, κοινωνικής κλπ. για κάποιες υποδομές. Άρα επίσης να αποθαρρύνουμε από επενδύσεις που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα. προσοχή όσον αφορά τις ασφάλειες και εγγύσεις. Πολλές φορές στην Ιταλία έχουμε ε, διευκόλυνση των δανείων που συνδέονται με το μισθό, αλλά αυτό οδηγεί σε ευξημένους κινδύνους. Εμείς θέλουμε να υπάρχει δεσμευτική μόγλευση. Αλλά όσον αφορά τα παράγωγα να προβλέψουμε αυτό το συντελεστή 3% για το κατόφλι. 12% επίσης για άλλες περιπτώσεις τραπεζικών δραστηριοτήτων. Κάλυψη της ρευστότητα, επιπλέον buffer για τις ε, τράπεζες που έχουν εκτεθεί όταν ε, ε διαπραγματεύονται τίτλους πιο ε, υψηλού κινδύνου. Τώρα για το... Για τώρα 507 θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να καταργηθούν οι εξαιρέσεις γιατί μπορεί να προέλθει από εδώ συστημικός κίνδυνος. Γιατί κάποιες τράπεζες έχουν πολλά κρατικά ομόλογα. για το CRD. Όπως και η πράσινη και η γκουε θέλουμε να έχουμε όριο όσον αφορά την, τις αμοιβέ του προσωπικού ανωτέρου και μέσου. Να υπάρχει εγγύηση για τον συστημικό κίνδυνο για να μην έχουν επομένω ιδιαίτερη, ιδιαίτερο κίνδυνο οι τράπεζες που έχουν εκτεθεί περισσότερο από άλλες. Αυτά είναι τα βασικά που θέλαμε να σας πούμε. Διαθέσιμος πάντα ο εισηγητής αλλά και οι σκιώδεις εισηγητές. Ελπίζουμε να προωθηθεί η πρόταση του Κοινοβουλίου για να βοηθηθεί η πραγματική οικονομία γιατί η Ευρωζώνη τώρα πρέπει να μπορέσει να τονώσει την ε, ζήτηση και δεν θα πρέπει να βάλουμε στενό κορσέ στις τράπεζες. Μάρκο Τζάνι. Ευχαριστώ και τον εισηγητή να ευχαριστήσουμε Πολύ λογική αρχική πρόταση και αφήνει περιθώρια για να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά σε κάποια σημεία που επιδέχονται συνεννοήσεις και επομένως εις βάθος να δούμε τι μπορεί να κάνουμε πάντως ξεκινάει με το δεξίο εισηγητής και θα υπάρξει με όλες τις πολιτικές ομάδες σε συνεργασία. Τώρα όσον αφορά τους γενικούς στόχους μας. Συμφωνώ βέβαια το ότι θα πρέπει το χρηματοοικονομικό και το τραπεζικό σύστημα να το κάνουμε πιο ανθεκτικό, πιο σταθερό και σε ετοιμότητα όχι μόνο για τυχόν κρίσεις, αλλά και να μπορούμε να τις προλάβουμε. Άρα, αυτό να κάνουμε, να χωθρογίσουμε τις τράπεζες και όχι να υπερβάλλουμε με μέτρα για το πώς θα προωθήσουμε εκ των υστέρων του αυτής της κρίσης. Αυτό θα πρέπει να είναι ο Μπούσουλας στη δουλειά μας. Επίσης, ένας άλλος στίχος με τον οποίο συμφωνούν και άλλοι συναδελφοί είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι το ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια νομοθεσία που βιαστικά θεσπίστηκε εν καιρό κρίσης. Να είναι όμως τελικά εύκολη στην εφαρμογή και, και κατανοητή. Αυτό είναι το καθήκον μας οποίων των κρίσεων. Να μπορούμε να έχουμε τέτοια νομοθεσία όπως σας είπα. Και ως προς τον κόσμο και ως προς τις τράπεζες και ως προς τις αρχές που καλούνται επί της νομοθεσίας αυτής είναι η βάση αυτή να λάβουν αποφάσεις. Ε, βέβαια, είναι περίπλοκη η ρύθμιση που πρέπει να γίνει, αλλά να βοηθά τις αποφάσεις. Τώρα, για τα πιο βασικά σημεία για την ομάδα μας είναι το θέμα του λόγου μόχλευσης. Και αυτό το συντελεστή. Θα πρέπει και αυτός να είναι απλός, θα πρέπει να είναι κατανοητός και να αποτελεί ένα κριτήριο ασφαλές όσον αφορά την υγεία μιας τράπεζας. Μετά τη μεγάλη κρίση του 2013 οι τράπεζες πασχίζουν να δουν πώς θα βρουν κάποιο υποκατάστατο για τον προβλεπόμενο δίκτυο ε, μόχλευσης γιατί απεδείχθη ότι αυτό που προβλεπόταν δεν ήταν αρκετό. Άρα για να βοηθήσουμε τις τράπεζες θα πρέπει να δούμε ε, πώς τι θα προβλέψουμε απλό, τι δεν θα έχει δαπάνες συμμόρφωσης γιατί τελικά οι τράπεζες μετακυλίουν αυτές τις δαπάνες στον τελικό χρήστη, τελικό καταναλωτή. Και βέβαια είναι το θέμα της πραγματικής οικονομίας, πολύ θετικά τα πώς τα βλέπει ο εισηγητής και εγώ θα ήθελα να κάνουμε ακόμα ένα βηματάκι, να μειώσουμε δηλαδή την απορρόφηση κεφαλαίων και να υπάρξει χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία, ε, να υπάρξουν κάποιο είδου ασφάλειες για τα νοικοκυριά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τονώσουμε τον, τον, τον, τον, τομέα των αγενήτων που ε, έχει πληγεί από κάποια κόπωση. Αυτά όσον αφορά δηλαδή τις ε, εμπράγματες ασφάλειας. Να καταλήξουμε σε μικρότερη έκθεση ή σε κινδύνους όσον αφορά αυτόν τον κλάδο, όσον αφορά τα ακίνητα. Ενδεικτικά σας λέω αυτά τα σημεία. Θα συνεργαστούμε με τους ε, συγκεκριτές ε, σκιώδης, τους σκιώδης και τον βασικό συγκριτή για να δούμε πώς θα κάνουμε πιο απλό το καθεστώς που διέπει μια πιο σταθερή τραπεζική πραγματικότητα. Και σε σχέση με αυτά που είπε ο πράσινος συνάδελφος Βαν δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε υπερβολικά τις μικρές τράπεζες. Αυτές δεν είναι συστημικός κίνδυνος. Να προσέξουμε βέβαια για ε, τη διασύνδεση αυτών των μικρών τραπεζών. Δεν αποτελούν μεν κίνδυνο, αλλά μια που είναι τόσο ε, στενά, τόσο πολλές συνδεδεμένες μεταξύ τους, ε, τελικά αποτελούν ένα συστημικό ρίσκο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Αυτό το τραπεζικό πακέτο είναι μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες αυτής της νομοθεσίας ούτως ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους, να ενισχύσουμε τη σταθερότητα αλλά και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως ό,τι αφορά αυτά τα διεθνή πρότυπα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε χωρίς όμως απλά να τα μεταφέρουμε στην Ευρώπη, χωρίς καμία κριτική σκέψη. Θέλω τώρα λοιπόν να σας αναφέρω κάποια σημεία, κυρίως ό,τι αφορά τους κινδύνους της αγοράς. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να εισάγουμε σε αυτό το πακέτο άλλους τομείς θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε τι εισάγεται σε αυτό το πακέτο και τι είναι αποτελεσματικό. Σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση, πιστεύω ότι το πακέτο αυτό είναι μια ευκαιρία να δούμε πόσο έχουμε προοδεύσει, να επιτρέψουμε στις εποπτικές αρχές να εξετάζουν τις θηγατρικές των τραπεζικών ιδρυμάτων και σε ό,τι αφορά την ρευστότητά τους. Η αναγνώριση της αρμοδιότητας της εποπτικής αρχής θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις συναλλαγές μεταξύ των Ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του αποθεματικού, σε ό,τι αφορά την εσωτερική ρευστότητα, είναι ανάγκη να εξετάσουμε το επίπεδο χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε για τη συμμετρία σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού για τις ανακεφαλαιώσεις θα πρέπει να διατηρήσουμε τη διαφορετικότητα των ιδρυμάτων δεν είμαι λοιπόν υπέρ μιας γενικής εξαίρεσης το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει αστάθεια τέλος ό,τι αφορά την αναλογικότητα συζητήθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αναλογικότητας. Η αλήθεια είναι ότι η αναλογικότητα στο ευρωπαϊκό σκηνικό είναι θετική, διότι υπάρχουν διαφορε... διαφορές. Από την άλλη όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να υπεραπλουστεύσουμε διάφορα πρότυπα ή και να επιτρέψουμε αυτή τη γενική απαγόρευση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εσωτερικά μοντέλα. Να αναπτύξουμε εσωτερικά μοντέλα, μάλλον, λαμβάνοντας υπόψη μας γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της αναλογικότητας. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητέ Το λόγο παίρνει ο εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Να αναφερθώ στο τελευταίο σχόλιο. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτόν τον φόβο ότι δηλαδή έχουμε πολύ χαλαρές απαιτήσει για τα ιδρύματα τα οποία θα ωφεληθούν από την αλογικότητα ειδικά στο NSF έχουμε μια αυστηρότερη ρύθμιση για τα μικρότερα ιδρύματα. Α, συγγνώμη. Ναι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι εφενός δίνουν λιγότερα δεδομένα, αλλά η αυστηρότερη ρύθμιση σημαίνει ότι έχουν μια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία. Είναι απλούστερα τα πράγματα αλλά βεβαίως ε, υπάρχει και η άλλη πτυχή. Οπότε η πρότασή μου το προβλέπει αυτό και οι προτάσεις που βλέπουμε από τον συνάδελφο Γκίγκολτ πηγαίνουν πολύ παραπέρα. Να έχουμε δηλαδή ειδικέ διατάξεις που θα είναι επιπρόσθετες προς τις άλλες για τα μικρότερα ιδρύματα για να μην ωφελούνται τα λάθος ιδρύματα. Εμείς λέμε ότι κανένα ε, ίδρυμα δεν θα μπορεί να ωφεληθεί ε, αν χρησιμοποιεί εσωτερικά μοντέλα. Εσωτερικά μοντέλα και αναλογικότητα αποκλείονται στην πρότασή μου, αποκλείονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις πάρα πολλές προτάσεις ε, που ακούστηκαν σήμερα για τις συνεισφορές. Η λοιπόν, η συζήτηση κατέδειξε το εξής απέχουμε σε κάποια πράγματα στις λεπτομέρειες, αλλά επί της αρχής ε, νομίζω ότι σε όλα τα σημεία για τα οποία μιλήσαμε σήμερα μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε ότι έχουμε ευρείες ε, πλειοψηφίες που οπωσδήποτε θα διαφέρουν ε, όσον αφορά τη σύνθεση αλλά οπωσδήποτε έχουμε μια καλή πιθανότητα να πάμε στο Συμβούλιο με μια ισχυρή διαπραγματευτική εντολή. Και νομίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να περάσουμε σε μια επικοδομητική έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και για την συζήτηση. Ευχαριστώ. Πράγματι ήταν μια επικοδομητική συζήτηση όπου όπως είπατε έχουμε διαφορετικές ευαισθησίες αλλά βλέπουμε και τις δυνατότητες λογικών συμβιβασμών οπότε εμένα με ενθαρρύνει αυτό όχι ότι είναι εύκολο αλλά είναι νομίζω κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να διεκπαιρεώσουμε επιτυχώς και να σεβαστούμε και το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι το εξή 7 ε, Μαΐου ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ μοιάζει μακριά αλλά δεν είναι τόσο μακριά αν σκεφτούμε και τον αριθμό των τροπολογιών Απαιτεί λοιπόν εντατική εργασία, συναντήσεις των σκιωδών, συζητήσεις. Ε, αλλά ξεκινάει αυτή η φάση σε μια καλή βάση. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εξέταση των κατεξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών μέτρων. Τρέχω στη πέμπτη τέτοια εξέταση. Είναι μια επιτυχής καινοτομία θα έλεγα και διαφάνεια και για την αποτελεσματικότητα του ρόλου μας στα σημαντικά αυτά νομοθετήματα που είναι οι πράξεις κατεξιοδότηση και τα εκτελεστικά μέτρα. Σήμερα λοιπόν η συζήτησή μας αφορά την τελική τεχνική συμβουλή για την αξιολόγηση ορισμένων στοιχείων ε, του κανονισμού του 2012 για το short selling. Μετά λοιπόν από αυτή την συμβουλή ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσουμε από την ΕΣΜΑ και την Κομισιόν ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα επανεξέτασης ε, του κανονισμού. και βεβαίως ε, καλώς ορίζουμε ακριβώ ε, τις απόψεις της Κομισιόν που προβλέπει η Κομισιόν για τα τρία σημεία, δηλαδή εξαίρεση από δραστηριότητες αγοράς, ε, μικρότερε απαγορεύσεις και διαφάνεια. και βεβαίως οι απαιτήσει δημοσιότητας και αποκάλυψή. Έχετε λάβει τα ενημερωτικά σημειώματα και όπως ξέρετε ολοκληρώθηκε το θέμα το 2011 με τον Πασκάλ Καμφέν, τον εισηγητή των Πρασίνων, οπότε τώρα αντιλαμβάνομαι ότι τα έχει αναλάβει ο Φιλίπ. Καλωσορίζω λοιπόν τους κύριους ε, Ρος και Μαρλούντερ από ΕΣΜΑ και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση και θα τους δώσω τον λόγο για να κάνουν μια σύντομη εισαγωγή Πέντε λεπτά ο καθένας, προτείνω να ακούσουμε πρώτα την ε, ΕΣΜΑ. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε να σας μιλήσουμε σήμερα όσον αφορά τις τεχνικές συμβουλές που είναι η έσμα όσον αφορά τον SSR. πούμε για την ευκαιρία να σας πούμε τις αρχές μας σκέψεις. Αυτό που σε εμπειρίες μας μέχρι σήμερα από την υποπτία και την εφαρμογή αυτού του τόσο απειρισμού οργανισμού, Η εντολή μας δόθηκε από την Κομισιόν τον Ιανουάριο πέρσι για τεχνική συμβουλή αυτών των θεμάτων του SSR που θα ισχύσει τον, τον Νοέμβριο. Και επομένως τον Δεκέμβριο, συγγνώμη, ο SSR άρχισε να ισχύει από 1η Νοεμβρίου 2012 και τελικά ε, υποβάλαμε τις πληροφορίες το Δεκέμβριο του 2017. Οπότε έχουμε πρώτα-πρώτα την απαλλαγή από κάποιες δραστηριότητε, δεύτερον την αυτή τη διαδικασία για βραχυπόδοσμους περιορισμούς και τη μέθοδο κοινοποίηση και αποκάλυψη των net short positions. Και επίσης είπαμε ότι θέλουμε τώρα να έχουμε περισσότερη διαφάνεια επίσης, να έχουμε καλύτερη υποπτία όσον αφορά τα όσα απαιτούνται βάσει του κανονισμού SSR και να μην μπορεί να παρακάμπτει κανείς τον κανονισμό Κάναμε επίσης κάποια έρευνα ε, στις αρχές να δούμε πώς στην πράξη εφαρμόζεται και όπως προείπα έγινε και κάποια δημόσια διαβούλευση. Πάντως ε, οι απαντήσεις ήταν ε, περιορισμένες μόλις 20 και λόγο αυτού του feedback και επειδή με το MIFID 2 που εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο Πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν σημεία που πρέπει να γίνει κάποιο είδου τροποποίηση, αναθεώρηση και άρα χρειάζονται οι σύμβουλες μας. Για παράδειγμα όσον αφορά το MIFID και MIFIR θα πρέπει να καταλάβουμε κάποια από τα ζητήματα που αναδύονται για πληροφορίες όσον αφορά την κοινοποίηση για τις συναλλαγές και επίσης την κατάρτιση κάποιου είδους μητρώου αρχείου για τις υποχρεώσεις που επιτάσσει το ΜΥΦΙΡ. Και επομένως όλα αυτά τα προωθούμε σε πρώτη φάση και ό,τι ερωτήσει είχαν σας απαντήσω τώρα όσον αφορά το πρώτο βασικό θέμα της εντολής η εξαίρεση για τις ε, δραστηριότητες αγοράς, market making, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική διαφοροποίηση σύμφωνα με το MIFID από τη μία μεριά και το τι προβλέπει ο SSR από την άλλη. Για τις market making activities on venue, οι market makers θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιο επιμελητήριο ή χώρο συναλλαγών εκεί που γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Και για συναλλαγές OTC δεν χρειάζεται κανείς να είναι μέλος. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι άλλα μέσα καλύπτονται όπως subscription right, convertible bond και εταιρικό χρέος. Επίσης νέο, ε, νέα απέτηση κοινοποίησης για τους market makers σαν κάποιους προειδοποίησεις αρμόδιες αρχές εκεί που υπάρχει μια θέση net short επί αρκετό χρόνο ούτως ώστε με καλύτερη εποπτεία της ε, επίκλησης της ε, εξαίρεσης. Επίσης να, πρέπει να τροποποιηθεί η διαδικασία κοινοποίησης ούτως ώστε μέσω της εξαίρεσης θα πάντα να είναι πιο ευέλικτα και ε, πιο απλή η διαχείριση από τις αρχές. Παρακατώ τώρα όσον αφορά το δεύτερο θέμα για τους βραχυπρόθεσμους περιορισμούς του Σόρσελινγκ. Εδώ έχουμε στοιχεία σοβαρά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και επίσης υπάρχει ασύμμετρη εφαρμογή στην Ένωση. Οπότε μια που το πεδίο εφαρμογή του βελνικέ είναι περιορισμένο θα πρέπει να γίνει εδώ αλλαγή από την απαγόρευση του ΣΟΣ selling θα πρέπει να είναι απαγόρευση όσον αφορά νέες θέσεις net short. Όχι πλήρης απαγόρευση, αλλά περιορισμός όσον αφορά την αύξηση της θέσης net short. Δεύτερον, επίσης έχουμε προτείνει μόνο η αρμόδια αρχή της ε, αμέσως σχετιζόμενης αγοράς από πλευράς ρευστότητος μπορεί να προωθήσει αυτή την απαγόρευση που είπαμε. Να μην μπορεί άλλη αρμοδιαρχή να επιβάλλει σύναφη απαγόρευση. Νομίζω αυτό είναι το πιο σωστό γιατί είναι μέσο, άμεσο και χρειάζεται αποτελεσματικότητα. Επίσης να περιοριστεί το βελνικές των ε, μέτρων όσον αφορά με μετοχικό κεφάλαιο όσον αφορά κρατικό χρέος ε, όταν αυτά είναι αντικείμενο συναλλαγών στην Ευρώπη σε ευρωπαϊκά τέλο πάντων χρηματιστήρια. Θα πρέπει επίσης όσον αφορά τη διαφάνεια για τα net short positions θα πρέπει τα κατόφλια να παραμείνουν για δημοσιότητα προς ε, τους μετόχους και 0,5 του εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, όποτε έχουμε υπέρβαση των κατοφλίων να έχουμε κοινοποίηση, όχι αργότερα από τις 3.30 των την επόμενη μέρα και η σχετική δημοσίευση μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Τέταρτον, κέντρο κατευθυνόμενο σύστημα κοινοποίησης και δημοσιότητος για υπολογισμό. Ε, στους ε, εμπλεκομένους. Αυτό θα δώσει περισσότερη διαφάνεια. Επίσης, υπολογισμός επί τη βάση του μετοχικού κεφαλαίου για τις net short positions όσον αφορά και επίσης και ενημέρωση του κοινού ε, ή των μετόχων. Επίσης να χρησιμοποιήσουμε το Legal Entity Identifier για νομικά πρόσωπα όταν γίνεται η κοινοποίηση των net short positions αυτών των νομικών προσώπων και επίσης να χρησιμοποιούμε την μέθοδο που ονομάζεται nominal ονομαστική, τον υπολογισμό των έξω, από όσον αφορά το κρατικό χρέο, όσον αφορά ε, και τα εργαλεία και τα, τα, τα, παράγωγα, αλλά και τα εργαλεία spot. Εν κατακλείδη, ευχαριστώ για την ενδιαφέρον σα και ό,τι ερωτήσει έχετε, να σα τι απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ, το λόγο έχει επιτροπή. Καλημέρα σε όλους. Θέλουμε βεβαίως να ευχαριστήσουμε την ΕΣΜΑ για αυτήν την λεπτομερή ανάλυση. Εξέτασαν όλα τα θέματα που ορίσαμε στην εντολή μας και πρωτίστως φυσικά τα κριτήρια των μελών για τις εξαιρέσεις. Διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον επίσης κάποια από τα εμπειρικά στοιχεία για τη χρήση του κανονισμού αυτού και βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί 46 φορές μόνο στην Ιταλία και στην Πορτογαλία μόνο για μετοχές και ποτέ για κρατικά χρέη που ήταν και βασικός στόχος αν θυμάμαι καλά του εργαλείου Πέρα λοιπόν από κάποιες τεχνικές ε, προσαρμογές που προτείνει η ΕΣΜΑ, η Επιτροπή θα εξετάσει την βασική χρήση του κανονισμού αυτού, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανησυχίες για τις οποίες δημιουργήθηκε. Σε τεχνικό επίπεδο τώρα, όπως ε, παρουσίασε η ΕΣΜΑ, λειτουργεί ιδιαίτερα καλά. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο όμως θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί δεν εφαρμόστηκε στον τομέα για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκε. Αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν θεωρώ ότι συμπεριλαμβάνεται στην αναφορά της, στην έκθεση της ΕΣΜΑ. Δεν κατακρίνω την έκθεση γιατί δεν ρωτήσαμε το συγκεκριμένο ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τα εργαλεία μετά που χρησιμοποιήθηκε ο κανονισμός αυτός. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα θα εξετάσουμε την τεχνική έκθεση. Είμαστε εκτός χρόνου όπως γνωρίζετε σε ό,τι αφορά το νομοθετικό ε, χρονοδιάγραμμα. Έχουμε μόλις 20 μήνες στη διάθεσή μας. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το προλάβουμε στην παρούσα θητεία της Κομισιόν. Θα εξετάσουμε όμως από κοινού μαζί με την ΕΣΜΑ κάποιες από τις τεχνικές προτάσεις βελτίωσης και την εφαρμογή, την τεχνική εφαρμογή των κανονισμών αυτών. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε ίσως να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κάποιος θα πρέπει να λάβει θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του το ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο α, κρίσης εθνικών χρεών. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει περάσει αρκετό χρόνος να πούμε ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατάφερε να αναχαιτήσει κάπως αυτήν την κρίση, μπορούμε να κρίνουμε και το συγκεκριμένο κανονισμό. Ο Φίλιπ έχει το λόγο. Ρομπέρτο, σε κοιτούσα όταν μιλούσε εκπρόσωπος της Κομισιόν γιατί αναρωτιόμουν διαβάζετε ποτέ τους Financial Times ή γενικότερα διαβάζετε ποτέ τον οικονομικό τύπο. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η οικονομική κρίση επιλύθηκε διαφορετικά. Βεβαίως λοιπόν δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ τον λόγο εργαλείο. Ίσως αν τα εξετάσουμε τα πράγματα θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ρεαλιστές, να μην είμαστε στη φούσκα μας και να έχουμε πραγματικές δοκιμές. Βεβαίως η πιο πραγματική δοκιμή θα ήταν αν προκύψει μια νέα κρίση. Αυτή τη στιγμή με την πολιτική που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα εργαλεία. Έχω μεγάλο σεβασμό για την Επιτροπή, αλλά πιστεύω ότι με αυτό το σχόλιο τους κάνετε να φαίνονται κάπως ανόητοι. Βεβαίως έχουμε πραγματικό ενδιαφέρον στον τομέα αυτό και καλωσορίζουμε τη δουλειά που έκανε η ΕΣΜΑ. Έχω μια ερώτηση όμως. Εξαιτία από τις, τις εφαρμογές του MIFID 2 θεωρείτε ότι πρέπει να εξετάσετε τις προτάσεις σας γενικώ. Ε, τι προτείνετε λοιπόν να μην κάνουμε τίποτα μέχρι να έχουμε μια αναθεώρηση ή αυτή ήταν μια γενικότερη ανακοίνωση ότι απλώς θα πρέπει να περιμένουμε επιμέρους ανάλυση από την υπηρεσία σας πριν προχωρήσουμε περαιτέρω από την ΕΣΜΑ. Πιστεύω ότι είμαστε ένα καλό σημείο να κάνουμε κάποιες προτάσεις και έχω μόνο δύο ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που κάνετε συμπεριλαμβανομένων προτάσεων που αφορούν κατευθυντήριες γραμμές και επιπλέον εντολές και θα ήθελα να έχω την οπτική της ε, Κομισιόν. Θα ήθελα να ξέρουμε ποιες είναι συγκεκριμένα οι προθέσεις της Κομισιόν δυνητικά ίσως θα μπορέσουν να έχουν μια ε, νομοθετική πρόταση. Κάποιες από τις προτάσεις της ΕΣΜΑ προϋποθέτουν ε, νομική εξέταση. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση της ΕΣΜΑ για την αλλαγή της, μακροπρο... της ε, απαγόρευσης. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή των συναλλαγών. Η ερωτήση μου λοιπόν είναι προς την Κομισιόν και προς την ΕΣΜΑ. Ευχαριστούμε. Ο Μάρκος Φέρμπε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Θεωρώ ότι με αυτά τα οποία είπατε επιβεβαίωσατε πως οι αγορές ανέμεναν την νομοθεσία μας και πλέον τα ομόλογα δεν επηρεάστηκαν όπως είπατε και εσείς. Αυτό νομίζω ότι βεβαίως δεν οφείλεται μόνο στην καλή μας νομοθεσία και όχι ακριβώς στην ρευστότητα που υπάρχει, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μετά από έξι χρόνια ένα θετικό απολογισμό του σχετικού κανονισμού. Οπότε δεν προβλέπεται νομίζω μια γενική αναθεώρησή του, αλλά μικρές μόνο τεχνικές προσαρμογές. Τι θυμάμαι και την συζήτηση που είχαμε κάνει τότε, που είχατε προβλέψει τον θάνατο της Δύσεως, ο οποίος τελικά δεν συνέβη. Επίση, η ΕΣΜΑ τονίζει στην έκθεσή τη ότι κατά τη χρονική στιγμή της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από εκθέσει συναλλαγών της MIFID 2 και ιδιαίτερα από τέτοιες συναλλαγές που αφορούσαν δραστηριότητες market making δεν ήταν ακόμα διαθέσιμες. Οπότε το ερώτημα μου είναι σε ποιο βαθμό η μη διαθεσιμότητα των στοιχείων αυτών επηρεάζει την ε, ισχύει και την εγκυρότητα των αναλύσεων. Θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά αν είχαμε τότε αυτά τα στοιχεία και ακόμα σε ποιο βαθμό άλλαξε η MIFID 2 την ε, δομή των ε, συναλλαγών σε σχέση με τις προτινόμενες ρυθμίσεις για τις βραχυπρόθεσμες απαγορεύσεις ε, του index trading, η, trading η ΕΣΜΑ προτείνει όταν υπάρχουν σοβαρά μικρές πτώσεις να μην ε, υπάρχει η δυνατότητα εμπορίας ε, των ε, επενδύσεων που ακολουθούς των τεχνών. Μήπως όμως εδώ πέρα δημιουργούμε ένα παραθυράκι μετά για τις ε, απαγορεύσεις για τα κρατικά <coughs> ομόλογα. Η ΕΣΜΑ προτείνει όπως όταν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες πτώσεις των τιμών να εξετάζονται σοβαρά για να μην καλύπτονται μόνο αυτές. Γιατί αυτή η πρόταση υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι τα τωρινά κατόφλια είναι πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά. Τι σημαίνει όντως ε, ε, σημαντική ε, πτώση της τιμής σε σχέση με μία απλώς σημαντική πτώση της τιμής. Τέλος, για την διαφάνεια προτείνεται ένα σύστημα για να ενέχουμε τις ακάλυπτες αγορές ε, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Ένα κεντρικό σύστημα ε, θα μπορούσε να μειώσει ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες στην αγορά τα ε, έξοδα και το διοικητικό βάρος. Ποιος είναι ο αρμόδιος, οι αρμόδιες αρχές θα πληρώνουν τέλη συμμετέχοντες στην αγορά. Τι αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Γκουαλτιέρη. Κύριε Καμάλ. Περίμενα εσείς να μιλήσετε πρώτα-πρώτα για τους σοσιαλδημοκράτες και αυτό ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πολύ ευγενικό αυτό. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η αμοιβαία υποχωρητικότητα. Όταν πρωτοβγήκε ο κανονισμός Μάρκος, δεν θέλαμε να το προχωρήσουμε και να το βάλουμε στο IFMD. Μετά κάναμε αυτόνομο κανονισμό για τα μη καλυπτόμενα CDS. Να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα με τα CDO και τα CDS. Και είχαμε προσκρούσει δυσκολίες. Και για όλα αυτά το θέμα ήταν τι θα γράφανε στον ισολογισμό οι τράπεζες. Πώς θα διαχειριζόντουσαν τις ζημίες από αυτά. Για να δούμε τώρα όμως εν προκειμένου τι έχουμε. Εμείς είμαστε υπέρ της πρότασης κομισιών και τόσο επί ΙΕΣ μας θέλουμε θετικά. Μας αρέσει το ότι προσέχετε το θέμα της ρευστότητας στην αγορά. Είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε η ΕΣΜΑ ότι δυστυχώς δεν είχε πολύ feedback από την διαβούλευση. Και επίσης εδώ όσο είπε ο Φίλιπ, ο Φίλιπ για Μίφιντ και Μίφιρ. της κοινοποίησης επίσης του 25-26 για το νέο καθεστώς Τώρα, έχω δύο ερωτήματα. Πόσο χρειάζεται για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις, πότε θα μπορέσουμε και τι άλλο. Τι άλλο θα βγει στην επιφάνεια. Πόσα ξέρουμε και πόσα δεν ξέρουμε δηλαδή από το σκηνικό αυτό. Άρα θα πρέπει να δούμε πρέπει να προσέξουμε αυτή τη διάκριση όπως ελεγχθεί για, το, για τους market makers. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε κίνητρα σε αυτούς για την παροχή υπηρεσιών. και να αναθεωρηθεί ο τη SSR, ώστε κάποιες δραστηριότητε να μπορούν να είναι OTC και να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η πρόβλεψη, η ρύθμιση για τις εξαιρέσει. Και τελικά μέχρι ποιου βαθμού τα παράγωγα και τα συναφή προϊόντα παραβλάπτουν την αγορά. Η απαγόρευση τελικά δεν συνδέεται αναγκαστικά με περισσότερη σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα. Πώς το βλέπετε. Γιατί πολλές φορές όταν μιλούν για μελλοντικά γεγονότα κάνουμε και λίγο την καφετζού. Οπότε θα πρέπει να δούμε σε σχέση με τι απαγορεύσει, αν θα είναι συναρμόδιε και άλλες εθνικές αρχές. Ποιε θα είναι οι απρόβλεπτε συνέπειε Μήπως θα έχουμε αποσταθεροποίηση στα χρηματιστήρια και γιατί ρευστούντα στην αγορά. Τι θα, ποιες θα είναι οι συνέπειες της ε, σύστασης σε σχέση με το ΜΥΦΙΡ υπάρχει πρόβλημα συμμόρφωσης. Για τη βαστή για την κοινοποίηση. Αλλά ενημερώνεται κάθε διετία ο SSR. Υπάρχει εδώ κάποια συμβατότητα, κάποια συνέπεια ή απλώς πρέπει να εξηγηθεί. Μπορούμε να κάνουμε κάποιε προσαρμογές και έτσι να υπάρχει με τον SSR συμμόρφωση και να αξιοποιηθεί η βάση δεδομένων και να υπάρχει για τις μετοχές τακτή πιο, πιο συχνή τέλο πάντων ενημέρωση έχει μπει ε, και κάποιο ε, χρονοδιάγραμμα από το 2020 για πέστε μου Μήπως κάτι δεν κατάλαβα. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. όχι. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε λάβει και Κάποιε ερωτήσεις. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο βεβαίω, αλλά το δικό μου το ερώτημα αφορά περισσότερο το κατόφλι και τον μηχανισμό διαφανείας. Έχετε λοιπόν αρκετές ερωτήσεις ε, για να απαντήσετε. Ποιος θα να ξεκινήσει η ΕΣΜΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις ε, και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω μία-μία. Ξεκινώντας, ε, στην ε, σύμβουλή μας ε, για την χρησιμότητα της βαρχιπρόθεσμης απαγόρευσης, λόγω της εντολής ακριβώς εστιάσαμε στην βαρχιπρόθεσμη μόνο. Δεν είπαμε τίποτα για την αποτελεσματικότητα μακροπρόθεσμων απαγορεύσεων και για να ολοκληρωθεί η εικόνα είχαμε και 12 μακροπρόθεσμες απαγορεύσεις από την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού από τρεις χώρες ε, που πάλι αφορούσαν μετοχές παρά οτιδήποτε άλλο. Απλά για να υπάρχει πλήρη εικόνα. Το 46 λοιπά αφορούσε βραχυπρόθεσμες απαγορεύσεις. Αυτό ως αφετηρία. Νομίζω επίσης ότι κάποιοι ενδιαφερθήκατε για το ότι με την ισχύ της ΜΥΦΙΤ ε, ίσως υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία ε, δεν θεωρούμε ότι θα αναθεωρούσαμε θεμελιωδώς τις συμβουλές μας. Ε, ε, είναι περισσότερο θέμα κάποιων αποχρώσεων που θα ωφελούνταν από αυτά τα δεδομένα. Οι περισσότερες συμβολές αφορά ακριβώς την λειτουργία του ίδιου του κανονισμού περί short selling και θα συνεχίσει να ισχύει θεωρούμε υπήρχε ένα ερώτημα για το τι μπορούμε να δούμε μετά την θέση ενισχύ της MIFID. Κατά βάση βλέπουμε ότι έχουμε πλέον πολύ περισσότερους που τα έχουν ενσωματώσει και είναι ήδη στο Μητρό και έχουν κοινοποιήσει τα σχετικά στις Εθνικές Αρχές ή την ΕΣΜΑ σε σχέση με 11 επί MIFID 1 έχουμε φτάσει τώρα σε 80-90 δεν έχουμε λάβει όλες τις κοινοποιήσεις ακόμα από τις εθνικές αρχές, αλλά οπωσδήποτε είναι ένας μεγαλύτερος αριθμός. Έτσι αλλάζει λοιπόν σε ένα βαθμό η δομή της αγοράς, αλλά σαφώς είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε τώρα για τον γενικότερο αντίκτυπο της εφαρμογής που έχει δύο μήνες προς ε, έξι εβδομάδες. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών για να φτάσουμε ε, στην βάση κάποιων δεδομένων, χωρίς αυτό να υποτιμά τις ε, συμβουλές που δώσαμε, γιατί θα έλεγα πως ε, τα περισσότερα από αυτά δεν θα επηρεαστούν. Θεωρώ ότι τα άλλα ζητήματα αφορούσαν δεν γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις ε, παράκαμψης, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε πως όταν θέλει να κάνει κανείς μία συμφωνία, σαφώς θα προσπαθήσει να βρει τον πιο βολικό τρόπο και βεβαίως εκθέσεις μέσω παραγόγων σε short sales είναι σαφώς ένας τρόπος να γίνει αυτό, γι' αυτό προτείνουμε να ευθυγραμμιστεί η βραχυπρόθεσμη απαγόρευση, ο ορισμός δηλαδή, με την μακροπρόθεσμη απαγόρευση. Δεν θα φορά τις άμεσες πωλήσει, αλλά την γενικότερη έννοια των καθαρών θέσεων short που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε την παράκαμψη μέσω παραγόγων. Μία άλλη ερώτηση αφορούσε νομίζω το κατόφλι για τα κρατικά ομόλογα. Εάν δείτε τον πίνακα 1 στη σελίδα 39 όπου εξετάζουμε τα κατόφλια και τα στοιχεία σημαντικών πτώσεων των τιμών που ίσως ε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια απαγόρευση βλέπουμε ότι για τις μετοχές είναι γύρω στο κατόφλι που υπάρχει ήδη γι' αυτό ζητάμε να μην αλλάξει προφανώς για ομόλογα έχουμε, δεν έχουμε ε, στοιχεία αυτή τη στιγμή γιατί καμία απαγόρευση δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πραγματικά στοιχεία, έχουμε κάποια εμπειρικά στοιχεία που έχουμε βάλει στην έκθεση που δείχνουν ξεκάθαρα ότι φαίνεται πως για κατ' καμόλογα ίσως να μην λειτουργήσει τόσο καλά το κατόφλι. Αυτό μπορούμε να πούμε, αλλά θα ήθελα να είμαι κάπως πιο επιφυλακτική για έναν κεντρικό μηχανισμό διαφάνειας που ανέφερε ο κύριος Φέρμπερ και τη χρηματοδότησή του είμαστε σκεμμένα επιφυλακτικοί και λέμε ότι θα μπορούσε να έχει κάποια πλέον ένα κεντρικό σύστημα, αλλά πράγματι υπάρχει το ζήτημα του ποιος θα πληρώνει, τι σημαίνει επιχειρησιακά η οικοδόμησή του. Ε, δηλαδή λέμε ότι θα μπορούσε να έχει κάποιο όφελος, αλλά πρέπει να το εξετάσουμε για να δούμε το πραγματική σχέση κόστους-οφέλους και το εάν οι εταιρείε θα ήταν διατεθειμένες να πληρώσουν κάτι τέτοιο του ότι βεβαίω θα σήμαινε για αυτούς ευκολία και λιγότερο κόστος για τις αναφορές. Για τα άλλα ερωτήματα. Γιατί θεωρούμε ότι ο ορισμός ε, μεταξύ short-selling και MIFID ε, θα πρέπει να παραμείνει ως ε, έχει. Νομίζουμε ότι τονίζεται και πάλι στην έκθεση ότι οι έννοιες είναι κάπως διαφορετικές γιατί και το εύρος του ορισμού στην Μύφιντ είναι πολύ μεγαλύτερο ενώ εδώ πέρα στον κανονισμό περί short selling αφορά την εξαίρεση για την απαγόρευση αυτή οπότε θεωρούμε ότι είναι διαφορετικός ο σκοπός και έχει νόημα να μείνει ως έχει. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Αν ξέχασα κάτι, πείτε μου. Ναι, ναι, να ρωτήσω λίγο για την ευθυγράμμιση. Πράγματι υπάρχει μια διαφορά αρκετά σημαντική ταυτόχρονα πρέπει να πω για τις μετοχές που εξαιρούνται έχουμε δυσκολία να λάβουμε τις πληροφορίες από εθνικές αρχές ακόμα και με το χρονικό πλαίσιο που έχουμε. Οπότε ας κάνουμε πρώτα σωστά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πριν ε, αποφασίσουμε να γίνεται συχνότερα. Αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε. Αλλά είναι νωρίς θα έλεγα ακόμα. Αλλά τελικά θα πρέπει να υπάρχει η σωστή διαφάνεια έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να μπορούν να το αντιμετωπίσουν το του δυνατόν. Μάλιστα πολλές ερωτήσεις ε, και για την Κομισιόν ε, και συγκεκριμένα ε, τι σχεδιάζετε να κάνετε. Εύκολη ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι. Να απαντήσω στο σχόλιο του Φίλιπ Λαμπέρτου ότι προσπαθούσα να πω με τα στατιστικά στοιχεία. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ενδιαφέροντα στο βαθμό που οι περιορισμοί στο άρθρο 23 εφαρμόζονται για μετοχές και σημαντικές πτώσεις στην τιμή με μετοχών. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση που βρίσκεται επίσης στην έκθεση της ΕΣΜΑ, σελίδα 101, είναι ότι έχουμε σημαντικές ε, παρατηρήσεις ε, του παραβίασης του κατοφλίου του 7% είχαμε 10% θα έλεγα που έφτασαν στο κατόφλι και εκεί πέρα οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αποφάσισαν να μην εφαρμόσουν την απαγόρευση αυτή και ακριβώ. εκεί είναι το θέμα. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρεια και μπορούμε να πούμε ότι μόλις ξεπερνούσαν το κατόφλι και αυξανόταν η απόδοση, δηλαδή έπεφτε η τιμή, αυτομάτως θα είχαμε απαγόρευση. Και εθνικέ αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να μην το κάνουν. Αυτό μια ενδιαφέρουσα εμπειρική παρατήρηση και νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για να δούμε γιατί δεν έχουν εφαρμόσει την απαγόρευση. Λέει στην έκθεση ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν το έχουν εφαρμόσει γιατί ήξεραν την αιτία και θεώρησαν ότι δεν ήταν αναγκαίο κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπήρχε νέα έκδοση ή κάποιο άλλο γεγονός στην αγορά που εξηγούσε την πτώση οπότε δεν χρησιμοποίησαν την απαγόρευση. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ερευνηθούν νομίζω σωστά πριν ε, καταλήξουμε σε μια άποψη. Και έτσι έρχομαι στο ερώτημά σας για το τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι είχαμε ακριβώ αυτή την εντολή γιατί μας ανησυχούσε η ρευστότητα, η εφαρμογή ε, και η διαφορετική εφαρμογή σε κράτη-μέλη της εξαίρεσης. Ε, καλωσορίζουμε το συμπέρασμα της ΕΣΜΑ ότι πρέπει να ωφεληθούμε από αυτήν, να ωφελείται κανείς εάν είναι μέλος μιας πλατφόρμας. Αν υπάρχουν δηλαδή διευθετήσεις market making με μια πλατφόρμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ωφελήσει από αυτήν την εξαίρεση γιατί αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για την ρευστότητα. Αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό με τρόπο σωστό χωρίς να υπάρξει κάποια νομοθετική διαδικασία που είναι δύσκολο για λόγους χρόνου. Θα συνεργαστούμε στενά με την ΕΣΜΑ επίσης. Αντιλαμβανόμαστε την πρόταση της ΕΣΜΑ πως εάν κάποιος είναι market maker και διατηρεί μια θέση short για πολύ καιρό δεν δημιουργεί πλέον αγορές, απλά διακρατεί μια θέση, οπότε τότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απέτηση κοινοποίηση για να έχουν μια γενική εικόνα οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές του τι συμβαίνει. Να εστιάσω τώρα σε αυτά τα δύο πράγματα να ξεκαθαρίσουμε την εξαίρεση για το market making και την σχετική δραστηριότητα να πούμε ότι είναι απαραίτητο να είναι κανείς μέλος σε μία πλατφόρμα αλλά μπορούμε να πούμε ότι αν αρχίσει να διακρατεί θέσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τότε πρέπει να το κοινοποιήσει. νομίζω ότι έτσι θα έχουμε μια ισορροπημένη βελτίωση του συστήματος ελπίζω να το πετύχουμε αυτό χωρίς νομοθετική αλλαγή γιατί δεν μπορώ να σας δώσω εγώ κάποια εγγύηση ότι το νομοθετικό πρόγραμμα της Κομισιόν που ούτως ή άλλως είναι πλήρες μέχρι το καλοκαίρι με πρωτοβουλίες για βιώσιμη, ε, βιώσιμα χρηματοοικονομικά και Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε και άλλο θέμα νομοθετικό. Το ρεαλιστικότερο είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτές τις διευκρινήσεις ε, και τις κοινοποιήσεις για μακροπρόθεσμες διακρατήσεις θέσεων στην ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς λέει ο Πρόεδρος. Οπότε, τώρα έχουμε καλύτερη εικόνα. Είναι σαφές ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία. Καταλάβαμε. Πάντως, κάποια πράγματα και θα Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε πώς προχωράτε το θέμα και θα ενημερωνόμαστε για τι θέση θα διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι θα γίνει, μήπως θα γίνει αλλαγή στην νομοθεσία ή θα χρησιμοποιηθεί κάτι άλλο με την ΕΣΜΑ. Φιλίπ, και εσύ θα συνεχίσεις να παρακολουθείς. Άρα είτε στην ομιλία πραγμάτευση είτε εδώ. Να δούμε τι αλλαγέ θα πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Εδώ τελειώνει η δουλειά που κράτησε τόσο πολύ. Η επόμενη η συνάντηση είναι τη Δευτέρα. Στις 3 η ώρα. Αλλά και